Allora. Care colleghe, e cari colleghi. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ ε, συνάδελφοι, καλημέρα. Χαιρετώ τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τη Κομισιόν που είναι μαζί μα στην ε, Ολομέλεια. Θα συζητήσουμε τις, ε, τα συμπεράσματα του εκτάκτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έλαβε χώρα από 17 έως 21 ε, Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 154 άρθρο 4 του κανονισμού συγκαλείται αυτή η έκτακτη σύνοδος ολομέλειας ε, για να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο για το σχέδιο ανάκαμψης και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση που διακόπηκε στις 10 Ιουλίου. Έχετε λάβει το πρόγραμμα των ψηφοφοριών με email. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε εγκρίνεται η μερίσια διάταξη και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Οπότε έχει καθοριστεί η ημερήσια διάταξη. Έχουμε τα πρακτικά της 8ης 9ης 10ης Ιουλίου 2020. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Κάποιες ανακοινώσεις. Οι αρμόδιες αρχές της ε, Γερμανίας μας κοινοποίησαν την εκλογή της κυρίας Μανουέλα Λίπα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς αντικατάσταση του κυρίου Κλάους Μπούχνερ. Η απόφαση ισχύει από 16 Ιουλίου 2020 μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19 Δεκεμβρίου 2019 λαμβανωμένης υπόψη της απόφασης της ε, Χούντα Electoral Σεντράλ του Ιανουαρίου 2020 και του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2020 το Κοινοβούλιο σημειώνει την εκλογή του κυρίου Φορ Ντισολέ ή Φεράντο με ισχύ από 3 Ιανουαρίου 2020 αντικαθιστά τον κύριο Γιουνκέρας ιδίως. Εύχομαι ε, λοιπόν καλή δουλειά και συμμετοχή στους νέους συναδέλφους. Η ομάδα των Πρασίνων μου ανακοίνωσε μια απόφαση τροποποίησης συμμετοχής στις κοινοβουλευτικές επιτροπές η οποία θα ισχύσει από τη στιγμή της ανακοίνωσής της. Ο κύριος Ρήπα θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ενέργειας και στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε. Λοιπόν, με την συζήτηση για τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν. Βλέπω όμως τον κύριο Βέμπερ που ζητάει το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν αρχίσουμε τη συζήτηση για την έκφαση και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θέλω να σας θέσω υπόψη κάτι κατεπήγον που είναι η κατάσταση στη Μεσόγειο. Είδαμε όλοι τις στρατιωτικές δράσεις από πλευράς Τουρκίας. Επίσης είδαμε τις αποφάσεις για την Αγία Σοφία που είναι ε, ένα παράδειγμα θρησκευτικού σοβινισμού. Ένα τέτοιο μνημείο ειρήνης και συμφιλίωσης, ένα σύμβολο, τώρα μετατρέπεται. Ε, αυτές είναι οι ε, τουρκικές ενέργειες και θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό το θέμα δεν είναι απλώς ελληνοτουρκικό ή κύπρο-τουρκικό, είναι ευρωτουρκικό. Και θα Θέλαμε να τονίσουμε παρουσία του κυρίου Μισελ και της κυρίας Φόντερ Λάιν ότι ε, συμπαραστεκόμαστε στους Έλληνες και Κύπριους φίλους μας. Βεβαίως παραμένουν ανοιχτή η διαβουλή επικοινωνίας και διαλόγου, αλλά έχει έρθει η ώρα να δράσουμε τώρα, να σκεφτούμε και κυρώσει κατά της Τουρκίας. Θα πρέπει να δράσουμε και να δράσουμε τώρα. Ήθελα να το θέσω υπόψη του σώματος. Σας ευχαριστώ κύριε Βέμπερ παρακαλώ τους ε, συναδέλφους που κάθονται στα έδρα να αναφορέσουν την ε, μάσκα όπως ορίζει ο κανονισμός. Λοιπόν, προβλέπεται τώρα η δήλωση του Συμβουλίου. Δίνω τον λόγο στον κύριο Μισελ για την παρέμβασή του. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Τέσσερα μερόνυχτα χρειάστηκε για να καταλήξουμε σε συμφωνία για πολύ περίπλοκα θέματα. Συμφωνήσαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πολιτή Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Και αυτή τη στιγμή ε, πιστεύω ακράδαντα ότι ε, ήταν ιστορική αυτή η συμφωνία. Δράσαμε άμεσα με ταχύτητα και σε λιγότερο από δύο μήνες καταλήξαμε σε μια συμφωνία πάνω από 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτή η αντίδραση είναι μαζική σε σχέση με το επίπεδο της οικονομίας και το μέγεθος της οικονομίας. Έχουμε μεγαλύτερη ε, ε, οικονομική συνεισφορά από τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Κίνα. Και μάλιστα η, η συμφωνία αυτή είναι πρωτοφανή από πολλέ από πολλές απόψει. Πρώτη φορά συμφωνήσαμε να δανειστούμε συλλογικά για να χρηματοδοτήσουμε δαπάνε. Και επίση είναι η πρώτη φορά που ε, τα δημοσιονομικά μας κονδύλια συνδέονται με τις περιβαλλοντικές μας φιλοδοξίες. Επίσης είναι η πρώτη φορά που ο προπολογισμό μας συνδέεται άμεσα με το κράτος δικαίου. Και είμαι πεπισμένος ότι η Ευρώπη ε, θα λάβει τέτοιες σημαντικές δράσεις. Και βρίσκομαι εδώ μπροστά σας με μία αναχείρα συμφωνία που επιτεύθηκε ομόφωνα 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έκαναν και υποχωρήσεις, έδωσαν και πήρα για να καταλήξουμε σε μια ισχυρή συμφωνία προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Μια συμφωνία που είναι ισορροπημένη και ορθολογική και γιατί, γιατί θα συμβάλλει στην υλοποίηση της ε, σύγκλησης, της ανθεκτικότητας και του μετασχηματισμού, της μεταρρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Next Generation EU, είναι ένα από τα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσει τη πανδημια covid COVID-19. Το συνολικό μέγεθο του Ταμείου ανάκαμψη είναι 750 δισεκατομμύρια ευρώ, 390 με τη μορφή επιχορηγήσεων και 360 δισεκατομμύρια με τη μορφή δανείων αποπληρωτέων. Και αυτά τα κονδύλια θα δρομολογηθούν προς τις περιοχές και τους κλάδους που επλήξαν περισσότερο. Και 30% των ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψη θα δρομολογηθούν για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγή. Και επίση τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψη θα πρέπει να πιάσουν τόπο και να συμβάλλουν ε, σε, σε μια χρηστή διακυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, θα προβλέψουμε 74 ε, τρισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα ε, θέλουμε με τα μέσα αυτά να καταβάλουμε προσπάθειες για να μειώσουμε τις ανισότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ε, ε, κατευθυνθούμε προς τη σύγκληση. Και σίγουρα ο πολιτή, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει κάποιες περικοπές και μερικοί στέκονται σε αυτές σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ στη διάρκεια της συζήτησης θα καλούσα να, δούμε το σημείο κίνησης, το σημείο αφετηρίας των διαφόρων πολιτικών. Και αν συγκρίνουμε με τη σημερινή κατάσταση, διαπιστώνουμε το, ότι το ΠΔΠ και το σχέδιο και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους μέτρα σε σχέση με τις δράσεις που έχουμε ήδη αναλάβει σε διάφορους τομείς, στον ψηφιακό, στον ορίζοντα Ευρώπη, στο έρασμος και τέλος προτείνουμε τη θέσπιση ειδικού αποθεματικού για το Brexit. Γιατί λαμβάνουμε υπόψη το γεγονό ε, ότι είτε με ή χωρί συμφωνία για το Brexit θα χρειαστεί οπωσδήποτε να στηρίξουμε τις χώρες και τους κλάδους που θα πληγούν περισσότερο από τις οικονομικές επιπτώσεις του Brexit. Και φυσικά υπάρχει ένα θέμα ε, που είναι ιδιαίτερα προσφυλές και συζητήθηκε ιδιαίτερα ε, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το θέμα των rebates, των επιστροφών που έμεινε ίδιο για μια χώρα και αυξήθηκαν οι επιστροφές για τέσσερις χώρες, είναι τμήμα τη συνολική συμφωνία δεδομένης αυτή τη πρωτοφανού κατάσταση, τη άνευ προηγουμένου κατάσταση και της ανάγκης να βρεθούν κονδύλια για το σχέδιο ανάκαμψη. Και, το... και νομίζω ότι αυτή η απόφαση για τα rebates είναι τμήμα τη συνολική συμφωνία. Επίση, για του ιδίου πόρου, είχαμε σφοδρέ συζητήσει και επίσημε και άτυπε για αυτό το κεντρικό θέμα, το θεμελιώδη ζήτημα, γιατί οι ίδιοι πόροι μπορούν να αποτελέσουν καμπή, για το μέλλον της Ευρώπης. Και νομίζω ότι μπορώ να δηλώσω ότι τα καταφέραμε, ακόμη και ε, πέραν αυτών που αναμέναμε πριν από λίγες εβδομάδες, γιατί δώσαμε κάποιο πολιτικό χρονοδιάγραμμα και επίσης αναδείξαμε με την εισαγωγή ενό ε, επιπλέον σημείου τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδείξαμε αυτήν την ιδέα ότι θα ξεκινήσουμε την ε, αποπληρωμή ε, του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ στην επόμενη φάση, που είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο στο πολιτικό επίπεδο, για να δεσμευτούμε όλοι, θα δεσμευτεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά θα δεσμευτούν και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Γιατί έχουμε κάποια μέτρα ε, πρόταση για τον ψηφιακό φόρο, για το φόρο αναπροσαρμογή το άνθρακα στα σύνορα, για το σύστημα εμπορία εκπομπών, για τα πλαστικά. Θα έχουμε λοιπόν περιθώριο για δημοκρατική πολιτική συζήτηση ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας με όλη την έννοια του όρου και θα έχουμε και συζητήσει στα εθνικά κοινοβούλια και είναι πολύ θετικό αυτό γιατί αυτέ οι συζητήσει για του ίδιου πόρου θα βρεθούν στο επίκεντρο των γενικών συζητήσεων για τον προσαρτορισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και φυσικά ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι θεμελιώδη. και σίγουρα θα το συζητήσετε και εδώ πέραν των όσων έχουμε προβλέψει σε θεσμικό επίπεδο για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού έργου, του νομοθετικού, του παρασκευαστικού έργου. Και ε, στα πλαίσια των Ταμείων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και, σε άλλα και για άλλα προγράμματα δαπανών στο άρθρο 11 των συμπερασμάτων ε, μιλούμε για επιμερισμό του πολιτικού ελέγχου μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια ε, του ελέγχου των δαπανών. Και σίγουρα οι συζητήσεις για το θέμα αυτό θα συνεχιστούν. Ένα άλλο θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφυλές και το συζητήσαμε. Ε, πάνε πέντε χρόνια που ανέλαβα που συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πρώτη φορά συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, για πρώτη φορά είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μία πολύ ε, μακροσκελή συζήτηση. Κατάματα μιλήσαμε ειλικρινά για τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Και φυσικά δεν καταλήξαμε κάπου, αλλά περάσαμε σε ένα σημαντικό στάδιο, πολύ ε, βασικό, γιατί προτείναμε αυτή την αιρεσιμότητα μεταξύ το οικονομικού σκέλους και του σκέλους της διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου. Και η κάθε θεσμικό όργανο θα αναλάβει το ρόλο του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα πλαίσια των ευθυνών να δώσει τις πολιτικές κατευθύνσεις. Όλοι θα πρέπει λοιπόν να επανερχόμαστε τακτικά σε αυτό το θέμα του κράτους δικαίου. Και αυτό το κεντρικό, θεμελιώδης, ζωτικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέλω να παραμείνει στο επίκεντρο της δημοκρατικής συζήτησης. Και θα ήθελα να καταλήξω στο εξή, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγε μέρες ξεπεράσαμε τους 600.000 θανάτους λόγω της πανδημίας COVID-19. Ε, η COVID-19 μας συντάραξε, μας κλώνησε, μας αναστάτωσε, τάραξε την, ε, τον τρόπο λειτουργίας των κρατών. Περιορίσαμε δραστικά τις θεμελιώδεις ε, και προσωπικές ελευθερίες. δοκιμάσαμε στιγνά την, ε, το υγειονομικό μας σύστημα. Θα πρέπει, διαπιστώσαμε, να είμαστε πιο δεσμευμένοι, πιο αλληλέγγυοι, πιο στιβαροί και φυσικά να έχουμε υπόψη την ανάγκη να επιδείξουμε ανθρωπιά. Η συμφωνία που σας παρουσιάζω σήμερα φυσικά είναι μια οικονομία που έχει κυρίως οικονομικές πτυχές, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί η συζήτηση που έχουμε σήμερα είναι η έννοια, το μέλλον, η κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη, στο μέλλον. Και νομίζω ότι γι' αυτό είναι ιστορική η συμφωνία και θα δείξω και κάποιο ρομαντισμό. Λόγω αυτής της πρωτοφανούς συμφωνίας θέλουμε και ένα πρόγραμμα στιβαρό για τους ίδιους πόρους, αποφασίσαμε να δανειστούμε από κοινού για να επενδύσουμε ε, στις προσπάθειές μας και να ανανεωθούμε την επόμενη τριακονταετία. Θέλουμε λοιπόν αυτή την Ευρωπαϊκή Ενότητα, αυτή διατρανώσαμε με τη συμφωνία αυτή περισσότερο από ποτέ. Και νομίζω ότι στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους Ευρωπαίους, μήνυμα εμπιστοσύνης, στιβαρότητας, σταθερότητας και το μήνυμα που δίνουμε στον κόσμο είναι ότι η Ευρώπη έδωσε το παρόν. Είναι εύρωστη, στιβαρή και όρθια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μισελ. Τον λόγο τώρα έχει η Πρόεδρος της ε, Κομισιόν, η κυρία Φοντερ Λάιν. Παρακαλώ. Εξακόσες χιλιάδες. 600.000 τα θύματα αυτού του φωνικού ιού. 600.000 ζωές χάθηκαν πρόωρα. 600.000 ε, ιστορίες που ε, γράφτηκαν μόνο μέχρι τη μέση. 600.000 οικογένειες σήμερα θρηνούν την απώλεια ενός μέλους τους. Και όλα αυτά θα παραμείνουν στη μνήμη τα μυαλά και στις καρδιές όλων μας και ξέρουμε ότι αυτό δεν έχει τελειώσει δυστυχώς. Όχι ακόμα. Και πίσω από αυτή τη θλιβερή πομπή βλέπουμε την τεράστια επίπτωση στις οικονομίες μας. Οι πολίτες μας, οι εργαζόμενοι μας, οι επιχειρήσεις μας. Όλοι υποφέρουν και όλοι αγωνίζονται. Η πανδημία αυτή μας έπληξε στην αρχή του έτους και όσο περνούσαν οι μέρες βλέπαμε να αυξάνονται οι ασθενείς και οι νεκροί. Και βλέπαμε την απειλή του διχασμού μεταξύ των κρατών μελών. Και ακούσαμε κριτικές ε, που μας πλήγωσαν, που μας δίχασαν, βορράς νότος, ανατολή δύση, συζητήσεις για ομόλογα κορονοϊού, που κατέληγαν με σφιγμένες γροθιές και τεταμένα δάχτυλα. Ήταν ζωφερή η κατάσταση και λίγες οι επιλογές. Και οι λίγες επιλογές που είχαμε επιτάπητος ήταν διακυβερνητικές. Δηλαδή εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, εκτός της κοινοτικής μεθόδου, εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θυμίζω επίσης δεν είχαμε συμφωνία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μας. Δύο χρόνια μετά την κατάθεση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια ευρωπαϊκή πρόταση για να αποφύγουμε τα αντανακλαστικά και τα σφάλματα του παρελθόντος. Μια ευρωπαϊκή πρόταση για μια ευρωπαϊκή ανάκαμψη. Το Next Generation EU αξιότιμοι ευρωβουλευτές, όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη ακόμα δεν έχει βγει από τις δυσκολίες. Αλλά τουλάχιστον βλέπει να χαράζει κάπου και να βγαίνει ένα φως. Αυτή την εβδομάδα ε, δεν παραμερίστηκαν μόνο κάποια ταμπού και ε, κάποιες ε, δρεωμένες αντιλήψεις, αλλά έγινε μια μεγάλη ε, καμπή 27 κράτη-μέλη υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δανειζόμαστε από τις κεφαλαιαγορές για να καταπολεμήσουμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση όλων των εποχών από κοινού. Το πρόγραμμα Next Generation EU είναι ένα μοναδικό, ένα ενιαίο εργαλείο ανάκαμψης με 750 δισεκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξουν όσους επλήγησαν σφοδρότερα. 750 δισεκατομμύρια ευρώ για να δώσουν όθηση στην ενιαία μας αγορά. 750 δισεκατομμύρια ευρώ για να επενδυθούν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την ψηφιοποίηση, ε, την αθεκτικότητα, τον εξυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής μας ενιαίας αγοράς. Βεβαίως, 27 κράτη-μέλη να συμφωνούν για ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους και τέτοιας μοναδικής η φύση χρειάζεται θάρρος, πολιτική βούληση, γιατί είναι πρόκληση. Και φυσικά κάτι θα δώσεις και κάτι θα πάρεις. Δεν είπαμε ποτέ ότι θα ήταν εύκολο. Αλλά πάντα αξίζει να αγωνίζεσαι για να επιτύχεις κάτι που αξίζει τον κόπο. Και θέλω να σε ευχαριστήσω, Σαλ, για την εξαιρετική συνεργασία και για την εμπιστοσύνη ε, για τη διαχείριση του Ταμείου. Και κοιτάξτε πόσο μακριά μας έφερε το αγωνιστικό πνεύμα της Ευρώπης. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που ορισμένοι έλεγαν ε, καθόλου επιχορηγήσεις μονοδάνεια». Σήμερα όμως έχουμε συμφωνία για 390 δισεκατομμύρια επιχορηγήσεις στο ταμείο αυτό, συν 360 ε, δισεκατομμύρια δάνεια. Βεβαίω, είναι λιγότερα τα δάνεια από εκείνα που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά κοιτάξτε από πού ξεκινήσαμε. Είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό. Και αρκετά σπουδαίο για να κάνει μια τεράστια πραγματικά διαφορά θα επενδύσει σε μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με ευρωπαϊκές προτεραιότητες και συνάδουν ε, με τις συστάσεις μας αναχώρα. Και ακριβώς επειδή αυτό είναι μια ευρωπαϊκή επένδυση, στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση είναι ουσιαστικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει εδώ πρωταγωνιστικό ρόλο. Ως συνομοθέτης, το Κοινοβούλιο θα έχει πλήρη λόγο στο σχεδιασμό της διευκόλυνσης και στη λειτουργία του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πλήρη διαφάνεια θα εξασφαλίσει τη λειτουργία. Είμαστε πρόθυμοι και για ένα διαρθρωμένο διάλογο για τις προτεραιότητες και για τις δαπάνες και για μια τακτική ανταλλαγή απόψεων ε, για τα εθνικά σχέδια και τη συνολική ε, υλοποίησή τους. Έτσι λοιπόν από κοινού μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα Next Generation EU θα πιάσει τόπο εκεί ακριβώς που χρειάζεται. Έτσι επίσης θα εξασφαλίσουμε ότι το Next Generation EU θα επιταχύνει ε, την ψηφιακή ανάπτυξη. Το 30% θα δαπανηθεί σε προγράμματα που συνδέονται με το κλίμα. Και αν ε, λειτουργήσουμε σωστά, είμαι πεπισμένη ότι το Next Generation EU θα κινητοποιήσει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις ανά τον κόσμο. Για να πάμε στο 5G, στις διάφορες νέες ε, τεχνολογίες, υποδομές, βιώσιμες μεταφορές, ε, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και ό,τι άλλο θέλετε. Και αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα καταπολεμάς την κλιματική αλλαγή και εξυγχρονίζεις. Θα υποστηριχθούν επίσης μεταρρυθμίσεις διαρθωτικές που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί. Και θα έχουμε και το Ταμείο δίκαιη Ανάκα, ε, Μετάβαση συγγνώμη, για να υποστηρίξουμε εκείνου ε, του τομεί και τι περιφέρειες που έχουν ακόμα μεγαλύτερα βήματα να κάνουν. Όπω γνωρίζετε, εγώ θα ήθελα περισσότερα. Αλλά η συμφωνία αυτή τη εβδομάδα εξασφαλίζει ε, αύξηση 125% για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που φτάνει στα 17,5 δις ευρώ πλέον. Και αυτό πραγματικά σημαίνει μεγάλη διαφορά επιτόπου. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Μέγας νικητής ε, της Συνόδου Κορυφής αυτής είναι οι νέοι ήδη Έχουμε πλέον ομόφωνη συμφωνία για την ανάγκη νέων ιδίων πόρων με σαφές χρονοδιάγραμμα. Και επίσης τους συνδέουμε τους ιδίους πόρους με την αποπληρωμή του χρέους. Αυτό είναι τεράστιο και ιστορικό άλμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέτει ε, τα θεμέλια για κάτι που πίεζαν εδώ και καιρό και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο πακέτο, μια δέσμη νέων ιδιοπόρων με ένα φόρο για τις ψηφιακές εταιρείε και ένα μηχανισμό προσαρμογής στα σύνορα για το διοξείδιο του άνθρακα και επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Θα πρέπει να τιμολογήσουμε το διοξίδιο του άνθρακα ε, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας στις χώρες μας και να αποφύγουμε διαρροή άνθρακα από άλλες χώρες για να παραμείνουμε και ανταγωνιστικοί αλλά και βιώσιμοι. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, επιτρέψτε μου να έρθω τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο βρίσκεται στην καρδιά την ίδια ε, την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι οι αξίες μας. Οι αξίες αυτές συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του κράτους δικαίου είναι τα ίδια τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές αυτές είναι και δεσμευτικές και πολύτιμες, ανεκτήμητες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύτηκε σαφώς να σέβεται το κράτος δικαίου και να προστατεύει τα οικονομικά μας συμφέροντα. Χαιρετίζω στεναρά αυτή την απόφαση και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε περισσότερα δημόσια κονδύλια από ό,τι στο παρελθόν με το πρόγραμμα Next Generation, αλλά με βάση αυτό τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει συνέχεια. Θα ξαναδούμε την πρότασή μας για το κράτος δικαίου του 2018. Θα συνεργαστούμε με τους συνομοθέτες για να διασφαλίσουμε ότι η πρόταση του 2018 προωθείται και όπου χρειάζεται βελτιώνεται. Η προστασία του προϋπολογισμού μας και ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι αλληλένδετα. Χέρι, χέρι και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προστατεύουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια ενισχύοντας την καταπολέμηση της απάτης με τους σωστούς ελέγχους και με μια βάση δεδομένων που να μας φέρνει σε θέση να γνωρίζουμε ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Και θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γίνει αυτό πραγματικότητα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρχισα λέγοντας ότι η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μας έδειξε το φως και μας έδωσε το φως στο τέλος του τούνελ. Αλλά όπου υπάρχει φως υπάρχει και σκιά. Και στην περίπτωση αυτή η σκιά είναι ένας πάρα πολύ πενιχρός, μακροχρόνιος ε, προϋπολογισμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ οδυνηρές αποφάσεις που ε, μας θλίβουν ε, που έχουν πολύ βασική σημασία. Σκέφτομαι εδώ το πρόγραμμα Horizon ή το πρόγραμμα για την υγεία, ουσιαστικότατο, ή το πρόγραμμα των επενδύσεων, InvestEU. Βεβαίως, αυξήθηκαν μεν όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά σε καμία περίπτωση όσο θα θέλαμε. Και εγώ πιστεύω ότι ε, το μέγεθος των εξωτερικών μας ιδιαίτερα ταμείων είναι πραγματικά ανησυχητικό. Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η αξία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη του κόστους. Βεβαίως καταφέραμε να αποφύγουμε ακόμα περισσότερες περικοπές όπως ήθελαν κάποια κράτη-μέλη. Αλλά το συγκεκριμένο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι δύσκολο να το καταπιούμε αυτό το χάπι και ξέρω ότι το κοινοβούλιο σας έχει την ίδια αίσθηση. Και πάλι εδώ, όμως, θα πρέπει να κάνουμε λίγο πίσω και να σκεφτούμε από πού ξεκινήσαμε. Ακόμα πριν ξεκινήσουμε καν, ο προϋπολογισμός αυτός είχε ένα έλλειμμα περίπου 70 δις ε, με το Brexit γιατί ε, μια μεγάλη χώρα ε, που συνεισέφερε δεν συνεισέφερε πια. Τα καλά νέα είναι ότι καταφέραμε περίπου να κλείσουμε όλο αυτό το έλλειμμα. Κάθε χώρα καλείται να πληρώσει περισσότερο. Και αν έρθει να προσθεθεί και το Next Generation EU, τώρα έχουμε μαζική δύναμη πυρός 1,83 13% περίπου του ΕΕΠ ολόκληρης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το PDP μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης ε, θα αυξήσει πάνω από 50% τις νέες σύγχρονες πολιτικές. Ρίξτε μια ματιά ανά τον κόσμο και πείτε μου ποιος άλλος μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο με μας. Κυρίες και κύριοι, τώρα έχουμε την ευκαιρία από κοινού να επιτύχουμε κάτι ιστορικό για την Ευρώπη η πίεση της κρίσης άνοιξε πόρτες που παρέμειναν ερμητικά κλειστές για πάρα πολλά χρόνια. Όσο θλιβερή και αν είναι η εφορμή, είναι και μια νέα ευκαιρία για την Ευρώπη, για την δική μας κοινότητα. Πριν από 10 χρόνια, στην κρίση του ευρώ και τη χρηματοπιστωτική, μπορεί να σώσαμε από τη διάλυση την Ένωση και το ευρώ αλλά το εσωτερικό μας τίμημα ήταν τεράστιο. Οι εθνικές μας οικονομίες ε, αναπτύχθηκαν αποκλίνουσες. Ε, Νέοι ναι, άνθρωποι ξενιτεύτηκαν, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν αλλιού δουλειά και μέλλον. Είχαμε πήρυψη ευθυνών, πολύ μεγαλύτερη μεταξύ των κρατών μελών. Και μέχρι σήμερα ε, είναι ορατές και αισθητέ οι ρογμές. Και αυτή τη στιγμή πράττουμε πολλά διαφορετικά και πιστεύω ε, αρκετά καλύτερα. 750 δισεκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεις κατά ε, Είναι ένα ε, σπουδαίο δείγμα αλληλεγγύης και επιθυμίας για μεταρρυθμίσεις. Αλλά το Next Generation σημαίνει πολύ περισσότερα από χρήματα. Στις προηγούμενες κρίσεις τα κράτη-μέλη και λόγω δυσπιστίας και καχυποψίας παρέκαμπταν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τότε σήμαινε αυτό μηδέν λόγο και μηδέν δυνατότητα ή διαμόρφωσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τούτη εδώ τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τούτη τη φορά ποντάρουμε στην κοινοτική λύση ε, και για το λόγο ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με μια ευφυή πρόταση έπεισε. Χάρη στο Next Generation EU όλα τα κράτη-μέλη μπορούν με τον ίδιο τρόπο να βοηθήσουν ε, τους πολίτες τους, τις επιχειρήσεις τους χωρίς ε, αυτό να στραγγαλίζει τους ε, κρατικούς προϋπολογισμούς. Και επειδή βασίζεται ακριβώς αυτή την κοινοτική μέθοδο, το Next Generation, ε, θα επουλώσει πληγές και θα μας φέρει πιο κοντά. Αυτή τη φορά θέτουμε την ευθύνη για τη μοίρα της Ευρώπης και τις ευκαιρίες για το μέλλον των παιδιών μας στους φαρδιούς όμως όλων μας. Είναι ένα βάρος που θα φέρουμε από κοινού με υπευθυνότητα και με υπερηφάνεια. Ζήτω η Ευρώπη. Στα γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο πρόεδρος ο κύριος Μάνφιντ Βέμπερ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, γεια όλοι. Κύριε Μισελ, κυρία Φόντερ Λάιν, αγαπητοί συνάδελφοι, η αλληλεγγύη επιστρέφει. Αυτό είναι το μήνυμα του Συμβουλίου. Τις τελευταίες αυτές μέρες είδαμε και την εναλλακτική, ένα σενάριο φρίκης ε, εθνικισμού και εγωισμού. Και εμείς ως ΕΛΚ είμαστε τώρα ιδιαίτερος ικανοποιημένοι για το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στέλνει ένα σαφές μήνυμα ενότητας. Πουθενά άλλου στον κόσμο 27 χώρες δεν δίνουν μια ενιαία απάντηση στην κρίση του κορονοϊού. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σαλ Μισελ, την κυρία Φοντελάιν την Αγγέλα Μέρκελ και τους δικούς μας διαπραγματευτές και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ε, πέρασαν πολλές άγρυπνες ε, ε, νύχτες, κάνατε καλή δουλειά και το ΕΛΚ σας στηρίζει στο πνεύμα αλληλεγγύης και ενότητας. Είμαι οπωσδήποτε ικανοποιημένες για την ε, συμφωνία, όχι όμως τόσο πολύ για το περιεχόμενό της, ε, γιατί βεβαίως είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, οπότε τώρα θα πρέπει να κριθεί το ζήτημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε γιατί ακούω τώρα διάφορα επιχειρήματα εδώ στους ε, διαδρόμους. Η πρώτη πρόταση του ΠΔΠ, το ανέφερε η κυρία Φοντερ Λάιεν, είχε κατατεθεί στο, είχε υποβληθεί στο Συμβούλιο το 2018. Οπότε μην μας μιλάτε τώρα για καθυστερήσει. Είχατε πάρα πολύ χρόνο. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι η τακτική διαδικασία τη σύμφωνη γνώμη με βάση την διαδικασία τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και ναι, έχουμε αρκετά σημεία κριτική. Αγαπητή Ούρσουλα, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι να καταπιούμε το χάπι το οποίο ανέφερε, ε, ειδικά στο ΠΔΠ. Στο ΠΔΠ θεωρούμε ότι δεν δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις στις προκλήσεις των επομένων 7 ετών. Πρέπει να είναι προσανατολισμένο προς το μέλλον και εγώ ως ερετός βουλευτής και πάλι δεσμεύομαι από τις υποσχέσεις που έδωσα στους ε, ψηφοφόρους μου. Υποσχέθηκε το ΕΛΚ παραδείγματος χάρη ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή, τώρα δεν υπάρχουν λεφτά. Το ΕΛΚ υποσχέθηκε ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τις μεγάλες ε, αρρώστιες όπως ο καρκίνος. Και τώρα δραματικές περικοπές στον προϋπολογισμό της υγείας. Σε καιρό κορονοϊού δηλαδή, είναι απίστευτο. Το ΕΛΚ υποσχέθηκε μια όθηση στην ευρωπαϊκή καινοτομία. Μόλις καθορίσει τον ε, στόχο 3% ε, του Συμβούλιο, χάνουμε έδαφος έναντι της Κίνας και της Ασίας. Και τώρα έχουμε περικοπές στο πρόγραμμα Horizon και το ΕΛΚ είχε επίσης υποσχεθεί ε, ισχυρή άμυνα, πολιτική γειτονία κτλ. Και, και τώρα και εκεί περικοπές και περικοπές και περικοπές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα μηχάνημα ανάληψης για τους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς. Έχει συγκεκριμένους στόχους. 90% των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Ταμείο New Generation EU θα πάνε απευθείας στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει πού ακριβώς θα ξοδευτούν αυτά τα λεφτά. Κάθε ηγέτης επέστρεψε στη χώρα του με έναν ωραίο φάκελο χρημάτων, αλλά υπάρχει μια ευρωπαϊκή λογική στο πώς θα ξοδευτούν τα λεφτά. Η αίσθηση μου είναι ότι θα ξοδευτούν από εδώ και από εκεί σε αυτούς που θέλει κάθε χώρα ο Γάλλος υπουργό είπε θα τα χρησιμοποιήσουμε σε κοινωνικό έργα, αλλού είπαν αυτοκινητόδρομους, αλλού είπαν θα μειώσουμε τους φόρους για να έχουμε ανάπτυξη. Και σε κάποιους μήνες θα είμαστε πάλι εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα παραπονιόμαστε ότι οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι ο σκοπός των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα παραπονιόμαστε ότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης. Αυτό το δράμα θα αντιμετωπίσουμε εάν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λεφτά για ευρωπαϊκά έργα όπως έκαναν οι προκάτοχοί μας με την Airbus παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να έχει συμφωνήσει παραδείγματος χάρη για ένα πραγματικό διεθνικό δίκτυο πέμπτης γενιάς για ένα σχέδιο για ενέργεια από το υδρογόνο, όπου θα μπορεί κάθε χώρα να χρησιμοποιεί τον εθνικό της φάκελο κατά τη διακριτική της ευχαίρεια. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε λόγο σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πού θα ξοδευτούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα φροντίζουμε να υπάρχει ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Και θα ήθελα να σα παρακαλέσω, πρόεδροι Μισελ και Φάντερ Λάιν, να προτείνετε 5-6 ευρωπαϊκά βιομηχανικά έργα και ενοτομία τα οποία θα δεσμευτούν τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν από τα χρήματα τομείων ανάκαμψη. Τρίτον, πρέπει να μιλήσουμε και πάλι για το κράτο δικαίου. Πρώτη φορά έχουμε σύνδεση των κονδυλίων με τον μηχανισμό κρατουσικαίου. Αλλά οι, πολίτες, οι ε, ηγέτες λένε διαφορετικά πράγματα. Ο Μακρόν λέει ότι υπάρχουν όροι, άλλοι ηγέτες λένε άλλα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κανόνες, ένα οδικό χάρτη. Να μην δίνονται χρήματα χωρίς να γίνονται σεβαστοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Και θα ήθελα και πάλι να ε, σας ευχαριστήσω για το αποτέλεσμα. Πρέπει να εργαστούμε τώρα σκληρά για μια γρήγορη λύση. Να εκμεταλλευτούμε τον καιρό που έχουμε μπροστά μας για να βρεθεί μια λύση για να βελτιώσουμε την συμφωνία αυτή. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βέμπερ. Τώρα, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Γκαρσία κυρία Πρόεδρε Φοντερ Λάιεν, κυρία Πρόεδρε Μισελ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με κάποια λόγια της Αρώ Λόπες, ε, ε, νοσοκόμο, που την περασμένη εβδομάδα στην κρατική κηδεία ε, που οργανώσαμε στην Ισπανία για τα θύματα του COVID, αυτά είπε. Δώσαμε ό,τι μπορούσαμε. Φτάσαμε στα όρια των δυνάμεών μας. Αντιληφθήκαμε περισσότερο από ποτέ γιατί επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα για να φροντίσουμε τον κόσμο, για να σώσουμε ζωές. Και παρόλο που κάποιοι σύντροφοί μας ε, θυσίασαν τη ζωή τους για αυτό το σκοπό, καλύψαμε τις ε, βασικές ε, και συναισθηματικέ ανάγκες των ασθενών και ήμασταν οι αγγελιοφόροι του τελευταίου αντίο για τα, για κάποιους ανθρώπους που πέθαναν μόνοι τους και άκουγαν από το τηλέφωνο μόνο τις φωνές των παιδιών τους. Κάναμε βιντεοκλήσεις, ε, κάναμε πολλά τηλέφωνα και χρειάστηκε να καταπιούμε πολλά δάκρυα. Αντιμετωπίσαμε τη χειρότερη κρίση τη γενιά μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αφήσει πίσω τι ε, τρέχουσε και τι επερχόμενε γενιέ. Η συμφωνία του Συμβουλίου, κυρία Φόντερ Λάιεν, κύριε Μισελ, θα περάσει στα στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης, οι... τα κράτη-μέλη συμφώνησαν για την έκδοση κοινού χρέους, ευρωπαϊκού χρέους, ευρωπαϊκού δανεισμού. Πριν από λίγου μήνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πρώτο αυτή την πρόταση και θα πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι ω θεσμικό όργανο γι' αυτό. Η απόρριψη των ε, αποφάσεων με ομοφωνία στη διακυβέρνηση των ευρωομολόγων είναι ένα επιπλέον ορόσημο που βάζει το φεδεραλιστικό στίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για δεκαετίες ε, είδαμε το μεταβέτο το πιο ζωφερό πρόσωπο της ακινησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα έχουμε μια ευκαιρία για να βρούμε ένα νέο τρόπο για τη λήψη αποφάσεων στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Σας ευχαριστώ για τις δεσμεύσεις που λάβατε και χάρη σε αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι διδάχτηκε από τα παθήματα της κρίσης του 2008. Και αν με την πολιτική λιτότητα αποφασίσαμε να σώσουμε τις τράπεζες και να αφήσουμε ουραγούς στους πολίτες, τώρα προτεραιότητά μας είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και αν θέλουμε να είναι προτεραιότητα, θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να καταφέρουμε μια κοινωνία πιο φιλοπεριβαλλοντική, πράσινη, πιο δίκαιη, πιο ψηφιακή. Η σοσιαλδημοκρατία δεν θα επιτρέψει η ανάκαμψη να επιβαρύνει μόνο τους πιο ευάλωτους μόνο αυτοί να επομιστούν οι ευθύνη. Γι' αυτό θα πετήσουμε έναν οδικό χάρτη με δεσμεύσει για του νέου ιδίου πόρου, για να μην στραγγαλίσουμε τα δημόσια εθνικά οικονομικά, ούτε την αγοραστική δύναμη των φορολογουμένων. Θα εξέλθουμε, αυτή την, θα εξέλθουμε από αυτή την κρίση μόνο με μια δίκαιη φορολογία. Γιατί είναι απαράδεκτο τα φορολογικά συστήματα κάποιων χωρών να επιτρέπουν στι πολυεθνικέ να εξοικονομούν εκατομμύρια ευρώ ει βάρο του της ευημερία μας και του κράτους πρόνοιας. Ο ιός συνεχίζει να μας χτυπά και γι' αυτό θα πρέπει η ανάκαμψη να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης όρισε θα διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψη και το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε επίγνωση τη ιστορική σημασία του Ταμείου Ανάκαμψη, αλλά δεν συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία σα για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι σοσιαλδημοκράτε δεν θα δεχθούν τι περικοπέ που προτείνονται στου μακροπρόθεσμου στόχου, που τη μια στιγμή σαν αυτή που ζούμε ε, είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε τη στρατηγική μα αυτονομία και να μειώσουμε τι διαφορέ και τι ανισότητε μεταξύ των κρατών μελών. Ελπίζουμε οι διαπραγματεύσει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό για να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση προγραμμάτων όπω Ορίζοντα 2020, το InvestEU, του LIFE, του Erasmus, του Ψηφιακή Ευρώπη, αλλά και του τους τομείς ε, συνεργασίας, αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν μπορούμε να αφήνουμε στη μοίρα του αυτού που μα χρειάζονται ε, περισσότερο που ζουν σε χειρότερε συνθήκε από εμά. Θέλουμε αλληλεγγύη εντό και εκτό των συνόρων μα. Και θα μείνουμε ακράδαντα προσιλωμένοι κατά οποιασδήποτε πρόταση που θα θέτει σε κίνδυνο το κράτο δικαίου. Γιατί το κράτο δικαίου και οι θεμελιώδει ε, αξίε ε, είναι το στίγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε ένα ευρώ δεν θέλουμε να δοθεί σε κυβερνήσει που δεν τηρούν το κράτο δικαίου και τι θεμελιώδει αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση συντρόφισσες και σύντροφοι. Όταν η πολιτική δεν είναι πια χρήσιμη για τους ανθρώπους, η κοινωνία δεν θα έχει πια εμπιστοσύνη στην πολιτική. Αυτή είναι η στιγμή για να εφαρμόσουμε την πολιτική με πι με μια πολιτική που συμφωνεί, που δεσμεύεται, που θέτει το κοινό συμφέρον ως υπέρτερο αγαθό, άνω των ατομικών συμφερόντων. Χθε μου είπε ένας νέος που ξαναβρήκα την εμπιστοσύνη μου ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε μια διαφορετική Ευρώπη. Στα χέρια μα ε, έχουμε κάτι τέτοιο. Α δεσμευτούμε για αυτού, για την Ευρώπη, για του πολίτε, άνδρε και γυναίκε. Για αυτού μια διαφορετική Ευρώπη είναι δυνατή. Σα ευχαριστώ κυρία Γκαρσία Πέρε. Τώρα για την ομάδα Renew, ο πρόεδρο Ντάτσεν Τσόλο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαν Μισελ, για την αποφασιστικότητά του να σφυριλατήσει ένα συμβιβασμό. Και επίσης, επειδή καλλιέργησες μια σχέση εμπιστοσύνης με το Κοινοβούλιο. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Σε λίγες μόνες εβδομάδες η Ευρώπη κατάφερε να δείξει μια πρωτόγνωρη αλληλεγγύη. Με ένα κοινό δάνειο που θα πρέπει από κοινού να αποπληρώσουμε για να ανταποκριθούμε σε μια από χειρότερες κρίσεις όλων των εποχών. Η ομάδα μου, Renew Europe, από τον Απρίλιο και τον Μάιο έχει κάνει παντιέρα της αυτό το σχέδιο ανάκαμψης και χαιρόμαστε που πλέον ε, γίνεται πραγματικότητα σήμερα. Είναι όμως ιστορική αυτή ε, η διάσταση αυτής της συμφωνίας ε, στο Συμβούλιο, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να μας εμποδίσει να συγκρίνουμε τα όσα έχουμε επιτάπητος με τις ίδιες μας τις φιλοδοξίες για την Ευρώπη το Συμβούλιο προτιμάει να ε, δώσει περισσότερα χρήματα σε εθνικά προγράμματα παρά σε κοινοτικά ε, προγράμματα. Αυτό δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη δική μας φιλοδοξία για μια στρατηγική επενδύσεων πραγματικά ευρωπαϊκή. Και αυτό το ευρωπαϊκό δάνειο που από κοινού θα αποπληρώσουμε δεν θα έχει νόημα εάν δεν χρηματοδοτήσουμε γνήσια ευρωπαϊκά προγράμματα. Και αυτό είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα εθνικά προγράμματα θα πρέπει να ενσωματώσουν αυτές τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και το Κοινοβούλιο ε, να έχει λόγο σε μια διοργανική συμφωνία για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Για να υπάρξει συμφωνία χρειάζεται ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο επαρκές για να μπορέσουμε να χρηματοδοτούμε τις πολιτικές του μέλλοντος. Ψηφιοποίηση, έρευνα, νεότητα, εράσμους, ε, το πρόγραμμα της υγείας ε, σε εποχές κρίσης είναι ένα από τα διδάγματα της κρίσης. Ε, δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την υγεία στον βωμό των επιστροφών, των rebates στα κράτη-μέλη. Ήδη πόροι. Επίσης, δεν θα είχε νόημα να δανειστούμε τόσα πολλά χρήματα αν δεν ξέρουμε πώς θα τα αποπληρώσουμε. Σαφής διοργανική συμφωνία και δέσμευση είναι απαραίτητη για να εγκριθούν οι ίδιοι οι πριν αρχίσουμε να αποπληρώνουμε τα δάνεια της ανάκαμψης. Αυτός είναι ο δικός μας όρος. Ένα πολύ ε, ακριβές χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να εγκριθεί πριν αρχίσει η αποπληρωμή. Τέλος η ομάδα μου θα συμφωνήσει μόνο εφόσον έχουμε ισχυρές εγγυήσεις για τη δυνατότητα να συνδεθεί ε, το Ταμείο Ανάκαμψης με το κράτος δικαίου. Όχι διακηρυκτικά, αλλά ουσιαστικά. Μόνο έτσι θα πιστέψουμε ότι αυτή τη φορά το έχουμε πετύχει. Θα έχουμε ένα νέο σύστημα με ε, σαφείς κανόνες που δεν στρέφονται κατά της Ουγγαρίας ή κατά της Πολωνίας ή κάποιο άλλου κράτους μέλους συγκεκριμένα, αλλά για να εγγυηθούμε ότι τα ευρωπαϊκά ε, χρήματα δεν χρηματοδοτούν ε, πολιτικούς που κάθε μέρα γεννούν την πλάτη στις θεμελιώδεις μας αξίες. Πρόεδρε, για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδειξε ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν περιορίζεται στο άθροισμα των εθνικών συμφερόντων όπου ο καθένας απειλεί με το βέτο θα κρυθούμε από τις κοινέ επιτυχίες και τις κοινέ αποτυχίες. Εδώ λοιπόν η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να είναι η ευκαιρία για να προσδιορίσουμε και να καθορίσουμε τη διακυβέρνηση για να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να ζήσουν τη μαγεία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος όπως τόσο τα είπατε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ομάδα ID ο κύριος Νικολαβή. Ιστορική μέρα για την Ευρώπη δήλωσε ο ε, Γάλλος πρόεδρος Μακρό έτσι, με πολύ ενθουσιασμό. Αλλά τα μεγάλα λόγια δεν σβήνουν ούτε τις μεγάλες αποτυχίες ούτε τις χαμένες ευκαιρίες. Το κοινό ψήφισμα που ε, καταθέτει κεντροδεξιά μέχρι την ακροαριστερά δεν αναφέρεται πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρέχει το Κοινοβούλιο μέσα σε 48 ώρες να ε, συνεδριάσει ε, και ευπηθώς να χαιρετήσει τη συμφωνία. Εμείς κομπάρσι είμαστε λοιπόν εδώ και ένα στούντιο μαγνητοφώνησης. Πού είναι η κοινοβουλευτική δουλειά και η νομοθετική. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να, για να γίνονται αυτά χρειάζεται κάποιο ελάχιστο χρόνο και νυφαλιότητα. Σήμερα γιατί βιάζεστε. Γιατί χάσαμε πολύ χρόνο εχθές. Πρώτα απ' όλα διότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ήταν μεγάλοι απόντες της ίδιας της υγειονομικής κρίσης. Η κρίση θα έπρεπε να είναι η ευκαιρία να επανεθεμελιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε γερά θεμέλια, υγιή, συνεργασία μεταξύ εθνών, ανεξάρτητη ε, βιομηχανία, τοπική κατανάλωση, χαμένη ευκαιρία, ύβρις, ε, ε, αμετροέπεια όλο πιο γρήγορα, όλο πιο ψηλά, φυγή προς τα εμπρός, χωρίς να μαθαίνουμε ποτέ από τα σφάλματα, απόντες από το συντονισμό απέναντι στην κρίση. Ε, και απούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί σήμερα να κάνει τα σφάλματά της και τα ελλείμματα να ξεχαστούν και θριαμβολογεί ε, Πολύ λίγα κράτη θα υποφεληθούν. 92 ώρες επίπονων διαπραγματεύσεων έδειξαν ότι τα εθνικά συμφέροντα πάντα θα έχουν το πάνω χέρι απέναντι στην φεδεραλιστική ουτοπία. Ναι κυρία Μέρκελ και κύριε Μακρόν, ακόμα αδράνεια ε, έχουν περικοπεί οι βοήθειες από 500 δις σε λιγότερο από 400 από τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων και εμπαρόδο μειώθηκε η ΚΑΠ, το Εράσμους και η έρευνα ποιο είναι ο βασικό στόχο, δογματικό και ιδεολογικό, παραμένει ένα ακόμα βήμα προ το ε, συγκεντρωτικό ευρωπαϊκό κράτο χάρη στην υπηρετική αμοιβιοποίηση του χρέου. Το ερώτημα είναι τι θα κερδίσουν τα έθνη μα, οι λαοί μα, πώ θα υποφεληθούν. Αυτή η οικονομική βοήθεια θα μπορούσε να αργωνωθεί με κάθε χώρα ξεχωριστά, η οποία θα έχει και το πλεονέκτημα να αποφασίζει τι θα κάνει και να μην τη θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ θα καταπιούμε αυτό το χάπι ε, που με καχυποψία ε, χαροπή ε, μας λέει ότι αυτό το, το τεράστιο χρέος το οποίο συνάπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά οφείλουν τα κράτη-μέλη θα το αποπληρώσουμε από τους ιδίους πόρους. Το ε, πρώτο βήμα για ένα ευρωπαϊκό φόρο. φόρο γκάφα, φόρο πλαστικό, φόρο για τον άνθρακα. Πολύ υποθετικά τα έσοδα και τελείως άγνωστα. Στην πράξη, οι εννέα χώρες που είναι καθαροί συνεισφορείς θα πληρώσουν τα σπασμένα ε, αυτού του νέου χρέους. Έτσι, για παράδειγμα, η Γαλλία θα έχει 40 δισεκατομμύρια από τα 750 και ε, θα αυξηθεί η συνεισφορά τη στην επόμενη εξέτεια. Αυτό είναι το ιστορικό για να ξαναπώ αυτά που είπε ο Μακρόν. Έναν πρόεδρο βλέπουμε να διαπραγματεύεται μια συμφωνία κατά του εθνικού του συμφέρον. Η, εθ... η υγειονομική κρίση δεν θα πρέπει να είναι η νέα πρόφαση για να συνεχίζει η ευρωπαϊκή οικοδόμηση όχι μόνο ερήμην των λαών αλλά και εις βάρος των θεμελιωδών του συμφερόντων. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους ο πρόεδρος Φιλίπ Λάμπερτς. Έχετε το... Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ονομάζονται Μαρκ Ρούτε, Ολλανδός Φιλελεύθερος, Σεμπάστιαν Κούρτς, Αυστριακός Χριστιανοδημοκράτης, Μέτε Φρέντριξεν, Σάνα Μαρίν και Στεφάν Λότβεν, σοσιαλιστές από τη Σκανδιναβία. Αυτοαποκαλούνται οι φιδωλοί. Εγώ θα έλεγα μάλλον οι τσιγκούνιδες. Γι' αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται σε μια αντλία χρήματος που οι χώρες του θεωρούν ότι τροφοδοτούν υπερβολικά. Απέναντι σε αυτή την προφορική, πρωτοφανή κρίση θα πρέπει να είναι απλώ αυτή η αντλία η Ευρωπαϊκή Ένωση μεσάζοντα μεταξύ των κρατών μελών που έχουν δυσκολίε και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Χωρί να βλέπουν ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε τεράστιε εντάσει στην ε, νομισματική ένωση και θα μπορούσε να αποβεί για την ύπαρξή τη. Αν ήταν έντιμοι όλοι αυτοί οι τσιγκούνιδε, θα εξηγούσαν στου συμπολίτε του πόσο έχουν υποφεληθεί οι χώρε του και συνεχίζουν να υποφελούνται από την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση. Οπότε είναι δίκαιο η συνεισφορά του στον ευρωπαϊκό προπολογισμό να είναι στο ύψο των ωφελών που απολαμβάνουν. Πολύ κοινικά όμω προτιμούν μόνο το ωφέλη τη Ένωση χωρί να καταβάλουν το απαραίτητο τίμημα. Ονομάζονται Βίκτορ Όρμπαν, χριστιανοδημοκράτη από την Ουγγρανία και Ταντέο Μοραβιέτσκι, Πολωνό συντηρητικό αυτοί ε, αποκαλούνται αντιφιλελεύθεροι. Εγώ θα έλεγα ψευδοδημοκράτε. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσημη αντλία χρημάτων που εξυπηρετεί το συμφέρον τη χώρα του, των ολιγαρχών του και των ιδίων. Αν ήταν όμω έντιμοι αυτοί οι ψευτοδημοκράτε, θα εξηγούσαν στου πολίτε του πόσο οι χώρε του επωφελήθηκαν και επωφελούνται ακόμη από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ότι ο σεβασμό των δεσμεύσεων που έλαβαν κατά την ένταξή του και κυρίω ο σεβασμό του κράτου δικαίου και των ελευθεριών είναι το αντίτιμο τη αλληλεγγύη. Με πολύ κινησμό όμω προτιμούν να τσεπώνουν τα χρήματα και τα ωφέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να περιμένουν να του χαμογελούμε και από πάνω. Αντίθετα όμω από όλου αυτού, μια πλειοψηφία αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα τη στιγμή. 200.000 Ευρωπαίοι έχασαν τη ζωή του ε, στην πανδημία COVID και οξύνθηκαν οι ανισότητε στην Ευρώπη εξαιτίας αυτής της κρίσης. Ε, περιορίζονται τα χρονικά όρια για να αντιμετωπίσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ. Η απέναντι στην Κίνα το Xi Jinping, το, Ηνωμένε Πολιτείε του Τραμπ, ε, τη Ρωσία του Πούτιν και, και την Τουρκία του Ερντογάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση μερικέ φορέ νιώθει μόνη τη να υπερασπίσει δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και έναν πολυμερή κόσμο και τάξη παγκόσμια. Ε, βέβαια, μερικές φορές η ομοφωνία έφερε τις 27 χώρες μέλη στο έλεος των πιο ακραίων. Βέβαια, οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακροτηριάστηκαν. Ήταν ήδη ανεπαρκή και ακροτηριάστηκαν κατά ένα τέταρτο, κυρίω για κάποιε πιο σημαντικέ κοινέ πρωτοβουλίε που θα εξυπηρετήσουν το μέλλον. Οι δημόσιες επενδύσεις χρειάζονται περισσότερα από ποτέ και παρόλα αυτά μειώσαμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και κυρίως ε, τη διάσταση τη φιλοπεριβαλλοντική της πράσινης ε, ε, συμφωνίας. Και αυτό φαίνεται στο Ταμείο Αγροτική ανάπτυξη, που είναι η πιο περιβαλλοντική πτυχή τη κοινή γεωργική πολιτική που περιορίστηκε στο μισό. Ε, πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα των κρουσμάτων όταν μειώνουμε τα προγράμματα έρευνα και δημόσιας υγείας και παρόλα αυτά εξαιτία του των τσιγκούνιδων μειώθηκαν αυτά τα κονδύλια. Βέβαια έχουμε και μια θετική πλευρά. Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το 30% των ευρωπαϊκών δαπανών για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Ελπίζουμε όμως να μην γίνει ένας καλοπισμός και να εφαρμοστούν εμπράκτος. Και χαιρετίζω τη συζήτηση ε, που μας αναφέρετε κύριε Σαλμισέλ. Ο μηχανισμός όμως ε, που είπατε για τους ιδίους πόρους ε, είναι το τυφλό σημείο και δεν είναι σίγουρο ότι θα εφαρμοστεί. Χάρη όμως την επιμονή της Άγγελα Μέρκελ και του Σαλμισέλ, το βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέμεινε αλόβητο. Και για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει συλλογικά με ένα κοινό δάνειο μαζικέ επενδύσει. Το θέμα τη αποπληρωμή, βέβαια, ένα άλλο τυφλό σημείο που έμεινε κρεμέ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, κατά τη γνώμη μου, ε, θα πρέπει επιτέλου τα κράτη-μέλη να χωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να εισπράττει φόρου. Κυρίω κατά των αρπακτικών πολυεθνικών, όχι μόνο του ψηφιακού τομέα, που ε, εφαρμόζουν, ε, εξοικονομούν εκατομμύρια και επίση έχουν δραστηριότητε που ρηπαίνουν το περιβάλλον. Ε, επίσης, χωρίς μια τέτοια έστω απαρχή δημοσιονομικής ένωσης, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι καταδικασμένη να μείνει ασήμαντη. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό η εκτέλεση αυτού του σχεδίου να ε, επαναφέρει το απαραίτητο αυτό στοιχείο στην επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εμπιστοσύνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επομιστεί πλήρως τις δημοσιονομικές του ευθύνε και θα δεχτεί αυτή τη χείρα που έτειναν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσει μέχρι να βρούμε ικανοποιητική συμφωνία ως προς τον όγκο των επενδύσεων, την κατεύθυνση, αλλά και το θέμα της αιρεσιμότητα με μοναδική πηξίδα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Και πριν ε, ολοκληρώσω, θα ήθελα να απευθυνθώ και πάλι στους συγκούνιδες και στους ψευδοδημοκράτες. Με τα λόγια και τα έργα τους που περιορίζουν και συρρυκνώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ε, οικονομικό χωνί, μια προσωποποίηση της ε, Σοβιετικής Ένωσης, ενσταλάζουν μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, το δηλητήριο του εθνικισμού στους συμπολίτε τους και ξεσηκώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες τους μεν κατά τον δε. Πριν από αυτούς, οι Βρετανοί συντηρητικοί ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο που γνωρίζουμε που οδηγεί. Αντίθετα, αντί να γυρίζουμε ένα στην πλάτη στον άλλον, εμείς οι Ευρωπαίοι περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να συσπηρωθούμε, να συνεργαστούμε και να εξασφαλίσουμε σε όλους σήμερα και στο μέλλον πιο αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης μαζί από κοινού θα βρούμε την ευφία και την δύναμη να χαράξουμε το δρόμο μας στον 21ο αιώνα. Αυτό είναι ο αγώνας μας και δεν πρόκειται να τον εγκαταλείψουμε ποτέ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ. Πριν συνεχίσουμε την συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει ο πρώτος γύρος ε, ψηφοφορίας στις τροπολογίες για την πρόταση ψηφίσματος για τα συμπεράσματα του εκτάκτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τις 10 και 30 μέχρι τις 11 και 45 η μέθοδος είναι αυτή την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει τις τελευταίες φορές άρχεται η ψηφοφορία έχετε μέχρι τις 11 και 45 τα αποτελέσματα θα τα έχουμε στις 13 και 30 ευχαριστώ κύριε Τσίλε παρακαλώ έχετε τον λόγο για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές κύριοι, αγαπητοί πρόεδροι, κυρίες και κύριοι πρόεδροι Κομισιόν και Συμβουλίου, το ECR έλεγε ότι έχει φτάσει η στιγμή να δράσει το Συμβούλιο. Τα κατάφερε τελικά. Δεν ήταν εύκολες οι αποφάσεις μετά από πολλές ημέρες διαπραγματεύσεων και το αποτέλεσμα βεβαίως περιέχει αρκετούς συμβιβασμούς και αρκετή ευελιξία. Τελικά όμως δείχνει πως υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός σε όλα τα κράτη-μέλη τα εθνοκράτη, κάτι το οποίο ε, μας ε, βοήθησε να καταλήξουμε σε μια λογική συμφωνία σαν αυτήν την οποία περιέγραψε ο Μάνφετ Βέμπερ. Υπάρχουν βεβαίω και άλλοι οι οποίοι διαφωνούν. Οι πολίτες στην Ευρώπη απευθύνονται κυρίως στις εθνικές του κυβερνήσει για να υπάρξει μια απάντηση στην πανδημία. Βεβαίω υπάρχει αλληλεγγύη, αλλά το ECR θεωρεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες μπορούν γρήγορα να δώσουν την απαραίτητη απάντηση. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν ε, ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να σώσουν τους ε, πολίτες τους και βεβαίως να χρησιμοποιήσουν μια αλληλεγγύη τους ε, πόρους με έλεγχο βεβαίως και ταυτόχρονα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα σημαντικότερα πράγματα είναι οι δουλειές, η ελπίδα για το μέλλον και εισόδημα βεβαίως για να επιβιώσουν. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου βεβαίως δεν είναι το τέλος της διαδικασίας και Είμαστε και εμείς επιφυλακτικοί στο ECR. Δεν θα δοθούν αμέσως τα χρήματα στις χώρες οι οποίες έχουν πληγεί άμεσα. Δεν θα είναι διαθέσιμα για 12 μήνες ή και ε, παραπάνω μετά από την δυσκολότερη περίοδο της πανδημίας. Ε, υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα ένας σαφής κίνδυνος ε, καθυστέρησης αντίδρασης στην κρίση σε μια δύσκολη στιγμή. Είμαστε έτοιμοι να επιφέρουμε τις απαραίτητες αλλαγέ με έναν επικοδομητικό τρόπο για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχουν βεβαίως κάποια ζητήματα που πρέπει να επιληθούν ειδικά στο ΠΔΠ. Λυπόμαστε για τις περικοπές στην γεωργία, την περιφερειακή ανάπτυξη που αφαιρούν χρήματα από την οικονομική ανάπτυξη, μείωση σε άλλα προγράμματα επίσης που στόχο είχαν ε, την ψηφιακή ατζέντα, την ανταγωνιστική εσωτερική αγορά και ζητήματα γεωπολιτικής ε, σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και Τέλος, ε, πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις για το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ όπου ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι σαφής. Δεν θα είναι εύκολο, είμαστε διχασμένοι ανακράτη-μέλη, αναπολιτικές απόψεις, αλλά δεν χρειάζεται να καθυστερήσει ε, άλλο η διαδικασία. Μπορούμε να οριστικοποιήσουμε αυτήν τη συμφωνία, η οποία είναι η καλύτερη δυνατή υπό τους όρους που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Ο πρόεδρος Μάρτιν Σίρντεβαν, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κυρία Φοντερ Λάιν, κύριε Μισελ, ε, δεν θα σας προξενήσει εντύπωση ότι δεν είμαι ιδιαίτερο ενθουσιώδης. Ε, τα κράτη-μέλη μετά από πολλά παζάρια επιτέλους ε, κατάφεραν να συνεννοηθούν, να αναλάβει, από... αναλάβει κοινά χρέη η Κομισιόν. Μέχρι εδώ καλά. Βεβαίω αναγκαστήκαμε να περιμένουμε πολύ για αυτό το σημάδι αλληλεγγύης. Η θέση μας ήταν πάντα σαφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει μια σαφή απάντηση στην, κρίση του κορονοϊού και να το συνδέσει με ένα στοιχείο αλληλεγγύης και ανάκαμψης της υπήρους μας. Λοιπόν, όταν τα συγκρίνουμε αυτά με την απόφαση του Συμβουλίου, τα πράγματα είναι απλώς απογοητευτικά. Έχουμε τώρα ένα μέσο το οποίο όχι μόνο υπολείπεται κατά πολύ του αναγκαίου όγκου για να αντιμετωπίσουμε μια κρίση η οποία σημαίνει ότι υπάρχει μια ύφεση κατά 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ αλλά έχουμε πάλι αντιπαραγωγικές επενδύσεις. Μια νοοτροπία η οποία θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πορεία, δυστυχώς δεν εμφανίστηκε πουθενά στο Συμβούλιο. Επικράτησαν οι εθνικοί εγωισμοί. Επίσης δεν υπάρχει κάποιος ρητός μηχανισμός για το κράτος δικαίου, για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ελεύθερο τύπο, ισότητα ανδρών και γυναικών, συνδικαλισμός. Αυτά δεν είναι αγαθά τα οποία ξεπουλούνται για λίγα δισεκατομμύρια. Είναι βασικά θεμέλια μιας δημοκρατίας και η αποπληρωμή των χρεών από τους ίδιους πόρους είναι επί της αρχής μια καλή ιδέα κυρία Φοντελάιεν αλλά βεβαίως με τον φόρο που έχετε προγραμματίσει τώρα 3 δισεκατομμύρια το έτος ε, και 390 δισεκατομμύρια δαπάνες αντιλαμβάνεστε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τώρα φορολογική δικαιοσύνη ένα ψηφιακό φόρο με υπολογιζόμενα ετήσια έσοδο 8 δισεκατομμύρια έναν φόρο 57 δισεκατομμυρίων ε, το έτος για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι επιχειρήσεις και οι υπερπλούσιοι πρέπει να πληρώσουν το μερίδιό τους. Τα είπατε κι εσείς ε, κύριε Φοντερλάιν. Κύριε Μισελ, αντί να μας κάνουν ε, μαθήματα οι Ολλανδοί που είναι φορολογικός παραδείσος, θα πρέπει επιτέλους να κλείσουν η φορολογική παράδοση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο αυτό δεν είναι αρκετά φιλόδοξο. Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις για το μέλλον. Δεν είναι σωστό να κόβουμε ακριβώς εκεί όπου χρειάζεται, δηλαδή στην ψηφιοποίηση, στην υγεία, στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και ταυτόχρονα να έχουμε στρατιωτικές δαπάνες οι οποίες αυξάνονται. Η Ευρώπη το Σαββατοκύριακο που πέρασε έχασε μια ευκαιρία και δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί μια δεύτερη τέτοια ευκαιρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Σίρτεβαν. Τώρα για τους μη εγγεγραμμένους ο κύριος Τζαρούσο για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και επί δεκαετίες η Ευρώπη προχωρούσε μειοπικά φτωχοποιούντας πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Εμείς ως Ιταλία ευχαριστούμε τον ε, κύριο Κόντε και βεβαίως ε, είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Το Next Generation EU σημαίνει ένα οριστικό τέλος στις πολιτικές εκείνες οι οποίες έκαναν διακρίσεις μεταξύ των πολιτών των διαφορετικών κρατών μελών. Γυρνάμε σελίδα. Βεβαίω χρειάζεται μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες των προγραμμάτων που πρέπει να ε, διορθωθούν. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα νέο υπόδειγμα για την Ευρώπη που θα έρθει μετά τον κορονοϊό. Μια αλληλεγγύη μεταξύ των, λατών, των λαών με ανάπτυξη και φροντίδα για το περιβάλλον. Δεν θα πρέπει ποτέ να γυρίσουμε προς τα πίσω. Στο πνεύμα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τους οποίους η Ευρώπη δεν θα υπήρχε. Σας ευχαριστώ. Μουρεσάν Σίγφριντ για δύο λεπτά. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, το μικρό θέλει να σας ευχαριστήσω τρεις φορές. Ε, δεν έχω πρόβλημα. ευχαριστώ. Ε, Καλωσορίζουμε και χαιρετίζουμε τη συμφωνία κύρια Φόντερ Λάιεν και κύριε Μισελ. Το μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σαφές. Χαιρόμαστε για τη φιλόδοξη υποστήριξη 750 δις για όσους έχουν πληγεί ε, πολίτες, επιχειρήσεις και περιφέρειες από τον κορονοϊό. Είναι πολύ σημαντικό τώρα να ε, τα σχεδιάσουμε σωστά αυτά πραγματικά για τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσο περισσότερα είναι τα κονδύλια τόσο μεγαλύτερος και καλύτερος πρέπει να είναι ο έλεγχος και ο δημοκρατικός με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον προπολογισμό για την επόμενη ετή περίοδο και αυτό πρέπει να γίνει σωστά γιατί είναι προπολογισμό για την Ένωση και μετά τον κορονοϊό ε, θα πρέπει να είναι επαρκής για να καλύψει ε, τις υποσχέσεις που έχουμε κάνει ε, στους Ευρωπαίους πολίτες. Είδαμε 27 ηγέτες να αγωνίζονται για 27 εθνικές προοπτικές. Τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αγωνιστική για την Ευρωπαϊκή Προοπτική. Ακούσαμε το Συμβούλιο, τώρα έχει έρθει η ώρα το Συμβούλιο να ακούσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποια είναι τα αιτήματά μας και τι θέλουμε να μπορούν περισσότεροι νέοι να ταξιδεύουν και να σπουδάζουν ε, αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γνωρίζουν πώς ζουν οι Ευρωπαίοι, ποιο είναι ο Ευρωπαϊκό τρόπο ζωή σε διάφορες χώρες ε, ενωμένοι στην Ένωση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο προπολογισμό για το Εράσμο. Θέλουμε να μπορούμε να χτίζουμε περισσότερα νοσοκομεία και να εξυγχρονίζουμε τα εφιστάμενα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την υγεία και μεγαλύτερη καινοτομία και έρευνα γι' αυτό προτεραιότητα στο ορίζον Ευρώπη. Δεν θέλουμε να μείνει κανείς ε, πίσω και ούτε στην άκρη στη δίκαιη μετάβαση. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερα κονδύλια το σχετικό ταμείο. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τον προπολογισμό της Ένωσης για την επόμενη επτάετη περίοδο. Πρόεδρε Φόντερ Λάιεν, είπατε ότι είναι πικρό χάπι προπολογισμό που πρέπει να καταπιούμε. Ε, όχι, δεν θέλουμε να το καταπιούμε έτσι. Να το διαπραγματευτούμε, να αρχίσουν διαπραγματεύσει και να τελειώσουν γρήγορα και να ψηφίσουμε γρήγορα. Διότι, κυρία Φόντερ Λάιεν, διατελέσατε υπουργό και εσεί, κύριε Μισελ, πρωθυπουργό και ξέρετε ότι το τελευταίο λόγο για το προπολογισμό τον έχει πάντα το Κοινοβούλιο. Γρήγορα να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είναι φιλόδοξος ο προπολογισμό μας για την επόμενη επταετία. Μποναφέη. Σιμώνα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτέλους, επιτέλους και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε ένα βήμα. Υπάρχει λοιπόν μια ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση του κορονοϊού. Μπορούμε για πρώτη φορά να μιλάμε για κοινό ευρωπαϊκό χρέος για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των οικονομιών μας. Νίκησε λοιπόν η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Έχασαν αυτοί που λέγανε ότι η Ευρώπη δεν χρησιμεύει σε τίποτα, ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει. Αυτοί οι οποίοι ήθελαν να επιστρέψουμε στα εθνικά συμφέροντα. Όλα αυτά ίσχυαν μέχρι που ήρθε ο κορονοϊός και προκάλεσε βεβαίως πάρα πολλές ζημιές στους ανθρώπους ε, κυρίως ε, που πέθαναν και υποφέρουν αλλά και σε αυτούς που έχασαν τις ε, δουλειές τους. Μάθαμε λοιπόν επίσης πως από την κρίση δεν θα βγούμε με το να υπερασπιζόμαστε ο καθένας την δική του χώρα αλλά μέσω ενός κοινού ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν κύριε Μισελ. Αν λοιπόν το Ταμείο ανάκαμψη είναι καλό, το ΠΔΠ χρειάζεται πολύ βελτίωση. Χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για να ανακάμψει η οικονομία μας. Δεν έχει νόημα να παρουσιάζουμε συνεχώς τέτοια σχέδια. Θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί στην διαδικασία αυτή. Και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στις νέες προτεραιότητες για το μέλλον, ξεκινώντας από το Green Deal. Οπωσδήποτε θέλουμε να δώσουμε αυτό το οποίο χρειάζονται οι επόμενες γενιές στην Ευρώπη με το πρόγραμμα Next Generation Group, με το πρόγραμμα ορίζοντα, με το Ταμείο δίκαιη Μετάβαση, το InvestEU για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, το Health for Europe για την υγεία, το Erasmus. Όλα αυτά όμως υφίστανται περικοπές και δεν μπορούμε να δεχτούμε να πηγαίνουν ευρωπαϊκά κονδύλια σε αυτούς οι οποίοι δεν σέβονται τις αξίες της, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Έχουμε κάνει λοιπόν κάποια σημαντικά βήματα, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλοι. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, κοιτάνε την Ευρώπη με εμπιστοσύνη και ελπίδα. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Γκαρικάνο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, Λουίς. Τα καταφέραμε πολύ και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρία Φαδερλάιν, και στο Συμβούλιο κύριε Σαλμισέλ. Εργαστήκαμε ακαταπώνητα για να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο ανάκαμψη φιλόδοξο για να μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει ενωμένη αυτή την κρίση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δύο ψηφίσματα τον Απρίλιο και τον Μάιο έδειξε το δρόμο και έδειξε ότι ήταν δυνατόν να καταλήξουμε σε συμφωνία, συνεργαστούμε. Ε, η Ευρώπη έκανε το καθήκον της τώρα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν το δικό τους καθήκον. Μερικέ χώρε ήδη γιορτάζουν σαν να κέρδισαν το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά ο δρόμο είναι ακόμη μακρύ μπροστά μα. Και αυτοί που θα λάβουν τα κονδύλια τίποτα δεν έκαναν ακόμη για να επιλύσουν τα προβλήματα που θα χρειαστεί να επιλύσουν. Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας λοιπόν. Θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε το χρόνο και την ευκαιρία για να πραγματοποιήσουμε τις αλλαγές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται η χώρα μας. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Ούτε τα 750 δισεκατομμύρια που θα χρησιμοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με κοινό χρέος και θα ε, πρέπει να το επομιστούν οι επόμενες, οι επερχόμενες γενιές καθήκον μα απέναντι στι μελλοντικέ γενιέ είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια για να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία. Μόνο με αυτό το σκοπό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια. Και αυτό το μήνυμα να το επαναλαμβάνουμε παντού, σε κάθε γωνιά τη Ευρώπη, σε κάθε γωνιά τη κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Να εξηγήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που καθυστέρησαν και τις επενδύσεις που θα πρέπει να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να κάνουμε μια πιο ανθρώπινη Ευρώπη, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τις ελευθερίες τους σε ένα καθαρό περιβάλλον, σε μια τεχνολογία που θα εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Και από το πώς θα δαπανίσουμε αυτά τα κονδύλια θα δούμε αν θα βγούμε αποδυναμωμένοι ή ενισχυμένοι από την κρίση. Είναι λοιπόν στιγμή ευθύνη και δέσμευση. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει το παν δυνατό ώστε αυτές οι σημαντικές επενδύσεις που θα κάνει η Ευρώπη να πιάσουν τόπο. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Καμπεμενώση. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Μισελ, κυρία φοντρελάιν. Λάιν. Η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά βεβαίω ε, πρέπει να πούμε κάτι για να μην ε, χάσει το νόημά της τα 27 τα χρόνια τα 20 τελευταία χρόνια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα κανόνων ακατανόητο για τους πολίτες μας και πριν από τον ε, κορονοϊό η Ευρώπη ήταν η περιοχή του κόσμου η οποία αναπτυσσόταν ε, το λιγότερο. Λοιπόν, το να μην γίνει η αυτοκριτική μας εδώ πέρα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί όπως είπαν αρκετοί Πράγματι έχει σημασία μακροοικονομική η συμφωνία η οποία επετεύχθη στο Συμβούλιο. Βεβαίως ακόμα δεν έχει καθοριστεί το πόσο θα ωφεληθεί η χώρα μου. Δεν ξέρουμε ε, πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι παρεμβάσεις και κάποιες από τις υποθέσεις που ακούγονται είναι ανισχυτικές γιατί από ό,τι φαίνεται θα τιμωρηθούν κάποιοι παραγωγικοί τομείς ε, της οικονομίας. Από την άλλη υπάρχουν ε, οι συστάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μου να περικόψει ε, συντάξεις ε, και κοινωνικές υπηρεσίες. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα βεβαίως, κόψαμε τις ε, συντάξεις ε, στην ε, Ιταλία για να χρηματοδοτήσουμε τα ηλεκτρικά πατίνια από την Κένα. Αυτή η υποκρισία λοιπόν από το Μάστριχτ μέχρι τη Λισαβόνα μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει γιατί ο κίνδυνος είναι ότι οι πολίτες θα αντιληφθούν ότι δεν έχετε αντιληφθεί την σοβαρότητα της ε, κρίσης και τα μέτρα τα οποία προτείνετε δεν είναι πανάκια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιδρούμε με κοινό ευρωπαϊκό δάνειο και επενδύσεις ε, σε μια οικονομική κρίση. Εμείς οι πράσινοι αυτό το κασορίζουμε. Αλλαγή υποδείγματος. Οικονομικά και πολιτικά είναι ευφύης λύση. Αν θέλουμε να βγούμε ενισχυμένοι από την κρίση χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το τίμημα όμως ήταν υψηλό για το βήμα αυτό. Εμείς θα λέγαμε υπερβολικά υψηλό. Για να δώσουμε τη συμφωνία μας. Εσείς μάλλον για να τη δώσετε κύριε Μισελ θυσιάσατε τον ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό ε, και εθνικά τώρα ε, θα δαπανηθούν τα κονδύλια. Το 2024 θα έχουμε πολύ χαμηλό προπολογισμό. αφού θα έχουν προηγηθεί λίγα χρόνια ευπορίας η ψηφιοποίηση, η προστασία της φύσης, άνθρωποι σε περιοχές ε, με ανθρακοριχεία, ε, ε, νέοι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το εράσμους πληρώνουν την ύφη και τα σπασμένα για άδικες επιστροφές σε αλαζόνες πρωθυπουργού. Πώς απαντάτε στην πανδημία με το πρόγραμμα EU Health. Το κάνετε περικοπές. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. 30% επενδύσεις λέτε για το κλίμα. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, πολλοί ε, έχουν αγωνιστεί και εδώ στο Κοινοβούλιο και στα κινήματα ε, για να τηρηθεί η Συμφωνία του Παρισιού. Δεν ισχύουν αυτά. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις για την κλιματική προστασία και για τη βιοπικιλότητα. Να εξασφαλίσουμε ότι κανένα πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα συγκρούεται με ε, το στόχο της Συμφωνίας του Παρισίου και να μην ε, χρηματοδοτούμε τους υδρογονάθρακες. Εμείς οι πράσινοι, ε, ντρεπόμαστε κύριε Μισελ, χρησιμοποιήσατε ως ατού διαπραγματευτικό το θέμα του κράτους δικαίου και υποχωρήσατε εκεί. Το κράτος δικαίου και η δημοκρατία θα πρέπει να είναι αυτονόητα στην Ένωση. Η Ένωση δεν είναι ένα ATM για την ανάληψη χρημάτων. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε ε, στο μέλλον τι θα κάνετε. Δεν μπορούν αυτά να οδηγηθούν σε εμπλοκή. Θα πρέπει να υπολογίζετε και να γνωρίζετε ότι θα υπάρξει αντίσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς είμαστε συνομοθέτες, δεν είμαστε στο θεωρείο των θεατών, των επισκεπτών. Θέλουμε συμφωνία, αλλά θα διαπραγματευτούμε και σκληρά. Γιατί ένα τόσο ε, τέτοιου ύψου προπολογισμό και με αυτού του όρου για μα είναι απλά απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριο Βανόβατφελτ. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία και πραγματικά ήταν οπωσδήποτε απαραίτητη. Ε, γιατί δεν, ναι, είναι πολυτέλεια για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τη στιγμή που ακόμα σοβεί ο κορονοϊός και η πανδημία με κοινωνικέ και οικονομικές επιπτώσεις να μην καταλήξουμε σε συμφωνία. Είναι τώρα ο απαραίτητο μοχλός στα κονδύλια αυτά για να επανέλθουν γρήγορα οι οικονομίες μας, να ανακάμψουν, αλλά... Ε, υπάρχουν και κάποιε ατέλειε. Το πρώτο αφορά ε, την αιρεσιμότητα. Ε, όπου προβλέπεται ένα φρένο έκτακτης ανάγκης. Αυτό τι είναι, ε, πώς θα λειτουργήσει, αν λειτουργήσει ε, και τι θα συμβεί σε περίπτωση αδιεξόδου σε αυτό το επίπεδο. Δεύτερο σημείο ασάφειας είναι τι γίνεται με την αποπληρωμή. Βλέπω διάφορες αρχές και κάπως το πλαίσιο το γενικό για το τι θα συμβεί, αλλά συγκεκριμένα αυτά πώς θα μεταφραστούν, ποιος θα το κάνει. Πρόκειται για 750 δισεκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή είναι τελείως θολά και αόριστα αυτά τα πράγματα. Και σίγουρα στο εγγύς μέλλον και στο απότερο θα υπάρξουν πολλές συμφωνίες. Έχω ακόμα ε, ερωτηματικά για τα ε, κριτήρια ε, έχουμε πραγματικά πολύ ψηλή ιστορικά ανεργία. Ε, τέλος πάντων, η συμφωνία κάνει περικοπές για τα ερευνητικά προγράμματα, για τα καινοτόμα προγράμματα. Μα ακριβώς αυτά χρειαζόμαστε για να είναι πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική η οικονομία μας. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Γκουσμάου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους ε, είναι σημαντικό προηγούμενο που δημιουργούμε. Αλλά μιλούμε για χρέος και αν δεν έχουμε ιδίους πόρους και αν δεν έχουμε κάποια πρόοδο σε αυτό, όπως δεν είχαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ουσιαστικά ε, προκαταλα... προκαταβάλουμε κονδύλια από μελλοντικού προπολογισμού. Και για χρέος μιλάμε, ας μην ξεγελάμε τους πολίτες μας. Και με αυτό το χρέος επανέρχεται και η περίφημη μακροοικονομική αιρεσιμότητα που έφερε μια ε, καταστροφική αντιμετώπιση της προηγούμενης κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταστροφική για την οικονομία, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και τους πολίτες. Και το τίμημα της ε, συμφωνίας αυτής είναι ένας πιο συρρυκνωμένος προϋπολογισμός. Ένας προϋπολογισμός που θα κάνει την Ένωση μια Ένωση ακόμη πιο άνισων χωρών. Θα την κάνει λιγότερη, πιο αποδυναμωμένη. Επίσης, θα χρειαστεί χρειάστηκε να εξαγοράσουμε τους, α, τις τέσσερις χώρες που αυτοαποκαλούνται φιδωλές που μιλούν για κανόνες αυτές οι χώρες αλλά δεν έχουν πρόβλημα να λαμβάνουν ε, πιο αυξημένες ε, επιστροφές στα περιθώρια του προϋπολογισμού. Μας κάνουν μαθήματα ηθικής αυτές οι τέσσερις φίδωλες χώρε στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέχτηκαν όμω αυτό τον εκβιασμό και τον εφάρμοσαν για να δώσουν τη συμφωνία τους στο σχέδιο ανάκαμψης. Μιλούν για κανόνες και ηθικοί οι χώρες αυτές, αλλά είναι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και μάλιστα παραβιάζουν συστηματικά εδώ και μία δεκαετία τους κανόνες για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, τουλάχιστον για η Ολλανδία και η Γερμανία. Οπότε προσυπογράφουμε αυτό το ψήφισμα, γιατί το ψήφισμα αυτό λέει με σαφήνεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα αποδεχθεί τον μακροπρόθεσμο προπολογισμό ως έχει. Γιατί ουσιαστικά θα οδηγήσουμε σε ακόμη πιο άνηση ένωση. Και έχουμε το σκάνδαλο αυτό των επιστροφών, των rebates, των επιταγών που δίνουμε στις πιο εύπορες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό θα πούμε στις μελλοντικέ συζητήσεις και όλες οι πολιτικές ομάδες ελπίζω να παραμείνουν πιστές στο περιεχόμενο του ψηφίσματος. Αρνούμαστε αυτό το δρόμο που μας οδηγεί σε μια πιο άδικη και μια πιο άνηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο ο κύριος Πουτσδεμόν. Σας ευχαριστώ. Τα νέα για τη συμφωνία το Σαββατοκύριακο αυτό ήταν πολύ θετικά και ελπιδοφόρα. Τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, η συμφωνία συνιστά πρόοδο. Αυτό περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα τα κράτη-μέλη θα αναδιανύμουν τους πόρους και ελπίζουμε να το κάνουμε αποτελεσματικότητα, με ευελιξία και κυρίως αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους. Γιατί τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από μεγάλες προσπάθειες που θα κινητοποιηθούν τα κονδύλια αυτά χάρη στο καταπληκτικό έργο που θα πρέπει να είναι η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλληλεγγύη. Αυτή είναι η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας μην το ξεχνούμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει ένα ισχυρό μηχανισμό ανάκαμψης, αλλά χάσαμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενέργεια για να υπηρετήσουμε και να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Ιδιαίτερα τους καιρού αυτού, που δραματικές ε, καταστάσεις όπως αυτών των, αυτής των Ουιγούρων ζητούν από, τους, ε, από την Ευρώπη να δείξει περισσότερο ηθικό παράστημα στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και χώρες που θα λάβουν αστρονομικά κονδύλια δεν θα νιώσουν την υποχρέωση να αντιμετωπίσουν διαφορετικά την αντιπολίτευση των εθνικών μειονοτήτων όπως γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς οι Καταλανοί. Η Ισπανία θα συνεχίζει να... Ε, συνεχίζει να δαπανά εκατομμύρια για να κατασκοπεύει τους ηγέτες της καταλανικής αντιπολίτευσης και τι θα κάνουμε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, νοείται οικονομική ανάκαμψη χωρί ε, δημοκρατική διάσταση. Ναι, στην Κίνα. Στην Ευρώπη όμω έχουμε την ευκαιρία να το αποτρέψουμε, γιατί είναι ένα εφιάλτη και δεν θα πρέπει να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Δελάγκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από τις τέσσερις ημέρες και νύχτες που περιέγραψε ο κύριος ε, Μισελ, ε, η συμφωνία αυτή ήταν ε, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Το καλό ήταν ότι έχουμε μια συμφωνία για έναν προϋπολογισμό και το πακέτο ανάκαμψης από τον ε, κορονοϊό και την οικονομική κρίση. Ε, βεβαίως ε, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να πω πως πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα... Δεν έχει τελειώσει ακόμα η υπόθεση. Ε, αυτό αφορά κυρίω ε, και το θέμα του κορονοϊού επειδή χιλιακάδα. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στα άσχημα. Περικόπτεται η χρηματοδότηση τη καινοτομία την οποία χρειαζόμαστε για να έχουμε ανάκαμψη, αλλά και το θέμα τη φύλαξη συνόρων, τη μετανάστευση. Στην προηγούμενη κρίση τη μεταναστευτική είπαν οι χώρε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι από κοινού, ευρωπαϊκά. Και λέμε θα έχουμε μια κοινή συνοριοφυλακή αυτό ακριβώς ο προπολογισμό περικόπτεται τώρα και ε, το γνωρίζω κύριε Μισελ πως στην επόμενη μεταναστευτική κρίση θα πείτε «Α, εδώ πέρα χρειάζεται μια ευρωπαϊκή προσέγγιση» και περνάμε στον άσχημο. Αυτό ε, το θέμα εδώ είναι το θέμα του κράτους δικαίου. Αλλά δεν έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Γι' αυτό εδώ πέρα εγώ θα πάρω, θα σφίξω το χέρι που μας απλώνει η κυρία Φόντερ Λάιεν στο θέμα αυτό και ακούγοντα βεβαίω το πόσο συμφωνούν οι συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση τη Πολωνία, τη Τσεχίας και τη Ουγγαρίας στα 27 κράτη-μέλη, πως το Ευρωπαϊκό, κράτο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει πολύ σοβαρά το κράτος δικαίου. Λοιπόν, τι είναι το σημαντικό εδώ πέρα. Προσθέτουμε ένα νέο στοιχείο, αλλά το θεμέλιο είναι ο σεβασμός για το κράτος δικαίου. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση αυτό το κείμενο τώρα που προέκυψε από το Συμβούλιο για να υπάρξει ανάκαμψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μαρκές για δύο λεπτά. Πρόεδρε, αυτή τη φορά έχουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση. Οι πολίτες, οι οικογένειες, οι επιχειρήσεις, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα κράτη-μέλη μπορούν να υπολογίζουν στην ευρωπαϊκή απάντηση. Αυτό περιμέναμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησε για την δημιουργία ενός Ταμείου ανάκαμψη και την κοινή ανάληψη ευθυνών. Η ευρωπαϊκή απάντηση στηρίζεται σε αυτό το Ταμείο και συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδειξε δημιουργικότητα και πρότεινε μια ισορροπημένη και φιλόδοξη πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και σε συνδυασμό με το σχέδιο ανάκαμψη. Τα κράτη-μέλη σίγουρα έμειναν ικανοποιημένα με τα οικονομικά κονδύλια που θα λάβουν. Αλλά έχουμε μία ανησυχία που, όπως είπε και η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμερίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ε, στο μέλλον θα έχουμε ε, κάποια στρατηγικά προγράμματα που θα αυξήσουν την ε, ανθεκτικότητά μας, όπως το έρασμο στο ορίζοντες Ευρώπη, ψηφιακή Ευρώπη, το EU for Health, η δημιουργική Ευρώπη, τα δικαιώματα και οι αξίες. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαίρεται για την ευρωπαϊκή ανταπόκριση, αλλά θα χρησιμοποιήσει κάθε μηχανισμό που έχει στη διάθεσή του για να καταλήξει σε ένα πιο στιβαρό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό υπολογίζουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το θεσμικό όργανο που μεριμνά για το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Μπορούμε όμως να υπολογίζουμε και στους ε, Ευρωπαίους ηγέτε που σε αυτές τι εκτενείς διαπραγματεύσει υπεράσπισαν περισσότερο το ευρωπαϊκό συμφέρον υπεράνω των εθνικών του συμφερόντων. Και ζητούμε και μία ενδιάμεση αξιολόγηση που θα αναλύει και το gender mainstreaming, τη συνεκτίμηση τη διάσταση του φύλου στι πολιτικέ και ε, θα μετρά και την πρόοδό μα σε σχέση με του κλιματικού μα στόχου. Θα πρέπει όμω κυρίω να συζητήσουμε τι πηγέ χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Θέλουμε ίδιου πόρου όπω το ψηφιακό φόρο ή το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το να στηρίζουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό αποκλειστικά ή σε μεγάλο βαθμό μόνο στο ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματο των κρατών μελών θα μα οδηγεί στι ίδιε διαμάχε και διενέξει κάθε 7 χρόνια. Και γι' αυτό η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, η κυρία Χάιερ, για δύο λεπτά. συντάραξε του Ευρωπαίου πολίτε απέναντι στην αδυναμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ οι οικονομίε μα, οι εργαζόμενοι μα έχουν πληγεί τα μάλα, ευθύνη μα είναι να του δώσουμε πάλι ελπίδα ελπίδα ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έστω και προσδόκητες οικονομικές κρίσεις για να γίνει ο κόσμος μας πιο πράσινος, πιο αλληλέγγυος, πιο ανθεκτικός, πιο καινοτόμος. Και με αυτό το πνεύμα έρχεται κρατών και κυβερνήσεων υιοθέτησαν το σχέδιο ανάκαμψης. Πρόκειται για μείζον επίτευγμα και πρόοδο για το μέλλον μας. Μια ιστορική στιγμή, αλλά πιστεύω ότι κανένα αυτό το κοινοβούλιο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, εκτό και αν είναι πραγματικά απόλυτα κακόπιστο. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σα απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια που καταλήξατε σε συμφωνία για αυτό τον έκτακτο προπολογισμό και σα στηρίζουμε με σθένο. Βέβαια δεν ήταν καθόλου εύκολο το έργο σα, αλλά ειλικρινά δεν ήταν αναμενόμενα κάτι τέτοιο. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν εγκλωβιστεί στην ομοφωνία και έχουν τι δικέ του δημοσιονομικέ περιορισμού που φέρνουν στην Ευρώπη, γιατί γνωρίζουν ότι θα κρυθούν αμήλικτα στι χώρε του. Αυτό όμω θα πρέπει να σταματήσει. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ε, στην, στο ψήφισμα που θα θετήσουμε σήμερα, εμείς οι Ευρωβουλευτές ζητούμε μία δέσμευση, σαφή και υποχρεωτική για την ταχεία θέσπιση νέων ιδίων πόρων. Όχι γενικού και όριστους όρου, όπω προκειμένου ή πιθανόν. Ζητούμε από του ψηφιακού κολοσσού που εφαρμόζουν τη φορολογική βελτιστοποίηση και από τι μεγάλε βιομηχανίε τη κίνα που ρηπαίνουν να, να αναλάβουν το χρέο, να αναβάνουν το βάρο αυτού του χρέου. Και αυτό είναι ο λόγο ύπαρξη ή πεντουσία αυτού του σχεδίου, να εξασφαλίσει την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών χωρί να επιβαρύνει περαιτέρω του Ευρωπαίου πολίτε. Θέλουμε ουσιαστικά να κατοχυρώσουμε σε νόμο αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Και το αίτημά μα εντάσσεται στη δυναμική της δικής σα συμφωνία, κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε από σήμερα να ξεκινήσουμε τις απαραγματεύσεις για αυτόν τον τακτικό προπολογισμό μαζί με εμπιστοσύνη, με φιλοδοξία και ταχύτητα. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Ο κύριο Μάντισον, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. κυρία Φαντελάιν, κύριε Μισελ. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, ε, να ακούω τον ενθουσιασμό που επικρατεί ε, επειδή επετεύχθη μια συμφωνία. Αλλά το πρόβλημα με μένα είναι οι λόγοι. Γιατί δανειζόμαστε από κοινού 750 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πραγματικός λόγος σύμφωνα με την Κομισιόν είναι ότι πολλά κράτη-μέλη δεν θα μπορούσαν να δανειστούν ε, υπ' αυτούς τους όρους από μόνα τους. Γιατί, γιατί ε, η οικονομία τους ε, δεν ε, λειτουργεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί, γιατί οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί έχουν εμποδίσει τόσο πολύ τα κρατη ώστε δεν λειτουργούν πλέον τα πράγματα. Δηλαδή τα κράτη-μέλη τα οποία ήταν πιο συντηρητικά, πιο φιδωλά με την οικονομική τους πολιτική όπως η Εστονία, η χώρα μου η οποία έχει το χαμηλότερο δημόσιο χρέος ε, στον κόσμο πρέπει να δεχτεί τον κοινό δανεισμό γιατί κάποια κράτη-μέλη ζουν πάνω από τα όρια τους εδώ και χρόνια. Και τώρα για το κράτος δικαίου. Δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε τις συνθήκες ε, γιατί οι συνθήκες ε, δεν θα επέτρεπαν ε, να δανειστεί η Κομισιόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν ξέρουμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτή την αποπληρωμή. Και είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα καταλήξουν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ελπίζω λοιπόν να βρεθεί ένα ευρωπαϊκό μόνο. Σας ευχαριστώ. Χαουτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα εγώ να απευθυνθώ στους πέντε φίδωλους ε, στο Συμβούλιο σας, όπου ε, όλες οι πολιτικές οικογένειες έχουν τα ζητήματά τους για να είμαστε δίκαιοι. Το ερώτημά μου λοιπόν προς αυτούς είναι τι σκέφτεστε πραγματικά. Δέκα χρόνια μετά την κρίση του ευρώ, όπου υπάρχει επι, επιτέλους μια όθηση για ένα σχέδιο δημοσίων επενδύσεων, να το περικόψουμε υγειονομική κρίση ας κόψουμε τον προϋπολογισμό της υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α κόψουμε τον προπολογισμό της έρευνα. Δηλαδή η επόμενη ε, κρίση θα είναι η κλιματική. Ας κόψουμε το Ταμείο της ε, Δίκαιης Μετάβασης. Ε, και παντού βεβαίως υποτιμάται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ας αναβάλουμε και πάλι το θέμα του κράτους δικαίου. Ναι εντάξει έχετε τις επιστροφές σας αλλά εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας δίνουμε την ευκαιρία το καλοκαίρι να ξανασκεφτείτε τις προτεραιότητές σας. Σας ευχαριστώ για 1,5 λεπτό Κύριο Ζόνσα. Σας... σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το σχέδιο ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης ε, ε, μας χρειάζονται. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που προετοίμασε το Συμβούλιο μετά από εκτενότατες διαπραγματεύσεις και με την συμμετοχή της Πολωνίας αξίζει αναγνώρισης και θα ήθελα να το τονίσω. Βλέπω ότι η ιδέα της αλληλεγγύης, της ευθύνη, της υπευθυνότητα, υπερίσχυσε των εθνικών εγωισμών. Γι' αυτό δώσαμε και εμεί τη μάχη μα. Και δεν θα πρέπει κανένας ε, να πληγεί από τη συμφωνία που είναι ο καρπός μιας τετραήμερης διαπραγμάτευσης. Και το θέμα της, του κράτους δικαίου φαίνεται εδώ. Η, Ουγγρανή, η Ουγγαρία, η Πολωνία είναι υπέρ του κράτους δικαίου, είναι υπέρ του καθαρού αέρα, υπέρ του καθαρού νερού. Ε, και δεν θα πρέπει με ψευδή και εσφαλμένα να κρυβεί μηνύματα να τιμωρήσουμε κάποιο έθνος ή κάποιο κράτος γι' αυτό και η αμεροληψία ε, είναι απαραίτητη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Θέλουμε ισοτιμία και αμερόληπτη εξέταση. Εμείς δεν φοβόμαστε τέτοια ανάλυση ε, για τα κράτος δικαίου. Δεν θέλουμε όμως να στηρίζονται σε ψευδείς δηλώσεις. Θέλουμε να απελευθερωθούν αυτά τα κονδύλια, να δρομολογηθούν στην αγορά, να φτάσουν στις περιοχές, στις επιχειρήσεις, σε εκείνους που χρειάζονται προστασία της θέσης εργασίας τους έχουμε νέα χρηματοδοτικά μέσα και έχουμε διάφορα στάδια και γι' αυτό χρειάζεται σημαντικός έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή. Αυτά και εύχομαι καλή επιτυχία στη χρησιμοποίηση των κονδυλίων στα κράτη-μέλη. Κύριε Σομαζέ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε. Ακούω ότι η συμφωνία που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ιστορική αλλά γνωρίζουμε από την εμπειρία μας και λόγω της διάβγειας μας ότι καμιά φορά οι ανοιχτές θύρες σφραγίζονται πολύ γρήγορα απέναντι στη λογική ε, της, ε, του ανταγωνισμού ε, θα το δείξει το μέλλον. Αλλά η ιστορικότητα δεν μπορεί να είναι βραχύβια. Η συμφωνία έγινε στο βωμό άλλων πολιτικών, ΚΑΠ, ε, πράσινη συμφωνία, υγεία, κοινωνικό ταμείο και έρευνα. Η συμφωνία επίσης έγινε με μια ανησυχητική επανεθνικοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Και πιστεύω ότι τελικά η συμφωνία αυτή τι δείχνει. Ότι τα εθνικά συμφέροντα κυριάρχησαν επί των ευρωπαϊκών πολιτικών που εμείς υποστηρίζουμε και προασπίζουμε για να κλείσω, θέλω να πω στο Συμβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο. Είμαστε συνομοθέτες και συναποφασίζουμε για την νομοθεσία και είμαστε και εγγυητέ της κοινοτική μεθόδου. Σας ευχαριστώ. Thank you. One minute, madam. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό, κυρία Αντινόλφη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τη 21 Ιουλίου γεννήθηκε η Ευρώπη της Αλληλεγγύης Οπωσδήποτε θα θυμόμαστε αυτή την ημερομηνία ως την αρχή μιας νέας εποχής 750 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταπολεμηθεί η οικονομική κρίση. Έχουμε έτσι ρίξει τον σπόρο της Ευρώπης ε, του μέλλοντος και οπωσδήποτε θα είμαστε γενναιόδοροι και θα δώσουμε και σε αυτούς ε, που δεν ήθελαν να περάσει αυτό το σχέδιο όπως οι Ιταλοί εθνικιστές και οι λοιποί. Και βεβαίω. Ε, οι χώρες οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται ως ε, φίδωλες ε, είναι απλά μειοπικές. Πώς είναι δυνατόν να περικόπτεται ο προπολογισμό υγείας εν το μέσο μιας υγειονομικής κρίσης. Πρέπει να ξαναξεκινήσει η ανάπτυξη ονότο της Ευρώπης ε, στον πολιτισμό, στον τουρισμό. Το όνειρο λοιπόν του Σπινέλη και των υπολείπων ίδρυτων ε, επιστρέφει για να σώσει την Ευρώπη η οποία μέχρι χτες ήταν η μηθανής. Πρέπει να προχωρήσουμε προς το εμπρός. Το μέλλον μας περιμένει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Κάσπαρη. Κύρια Πρόεδρε, συγχαρητήρια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για αυτήν την γρήγορη συμφωνία. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα, ένα μήνυμα για το ότι η Ευρώπη παλεύει, το, για το ότι έχει διαφορετικά συμφέροντα, αλλά τα κράτη-μέλη είναι τελικά σε θέση να καταλήξουν σε κάποιε κοινέ θέσει. Και αυτό είναι σημαντικό για του πολίτε. Μπορούμε να βασιστούμε στην Ευρώπη, υπάρχει αλληλεγγύη. Ε, είναι αυτό το έγγραφο βεβαίως μια καλή διαπραγματευτική βάση, αλλά δεν θέλουμε απλά να το δεχτούμε έτσι. Τα λεφτά θα ξεκινήσουν να ρέουν ε, από πρώτη πρώτου. Έχουμε λίγο καιρό μπροστά μα. Έχουμε λοιπόν κάποια πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Έχουμε κάνει αρκετά για να διασφαλίσουμε ότι τα λεφτά θα πάνε προ λογικέ επενδύσει και όχι στο να διατηρήσουν ξεπερασμένες δομές εν ζωή. Γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκός προγραμματισμός όπως κάνουμε ήδη στα διαρθρωτικά ταμεία. Γιατί επέμειναν τα κράτη-μέλη να έχουν δικά τους προγράμματα. Η δεύτερη μου ερώτηση ε, προς εσάς κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου είναι η εξής. Πώς θα διασφαλίσετε το ότι δεν θα έχουμε μόνο το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ή 2-3 τα επόμενα έτη, αλλά το 49% το οποίο ξοδεύουν τα κράτη-μέλη του ΑΕΠ να χρησιμοποιείται σωστά. Γιατί βεβαίως μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αποτελεσματική μόνο εάν τα κράτη-μέλη λάβουν τα σωστά μέτρα με το 49% του ΑΕΠ που διαθέτουν εκείνα. Είναι ξεκάθαρη λοιπόν η προσδοκία που έχουμε από τα κυβερνήσει και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Βέλκεν. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Φοντερ Λάιεν, κύριε Μισελ, είναι θετικό το ότι προέκυψε ένα αποτέλεσμα από την διαπραγμάτευση. Δεν είναι καλό συμβιβασμό όμω. Το πικρό χάπι το οποίο αναφέρατε σήμερα δεν θα το καταπιούμε έτσι απλά η πρότασή σας ε, κόβει ε, από τα πράγματα που είναι σημαντικά για το μέλλον. Το InvestEU, το πρόγραμμα για το κλίμα. Περικόπτεται πάρα πολύ. Για την ε, δίκαιη κοινωνική μετάβαση από τα 40 περιεκόπηκε το σχετικό πρόγραμμα στα 17 δισεκατομμύρια. Περικόπτεται την πολιτική της συνοχής σε 42 εκατομμύρια το έτος. Μιλάμε για Next Generation EU, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, την υγεία. Πρέπει όμως να ασχοληθεί με την επόμενη γενιά, όχι με εμάς. Είναι λοιπόν απαράδεκτο και το να παραμελούμε αυτές τις προτεραιότητες των πολιτών ε, δεν είναι σωστό. Πρέπει άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει δικαίωμα λόγου για να το εμποδίσει αυτό. Μετά έρχομαι στο αδύνατο σημείο. Το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου είναι το κοινό θεμέλιο της συνεργασίας ε, και είναι και η ομπρέλα που προστατεύει τα δικαιώματα μας. Γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο πικρό αυτό το χάπι. Εμείς θέλαμε πραγματικά να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός κράτους δικαίου για να νιώθουν ασφαλείς ε, οι δημοσιογράφοι, οι διαδηλωτέ, οι δικαστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτό, Κέρνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Φόντερ Λάιεν, κύριε Μισελ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Είναι καλό που βγήκε ένα αποτέλεσμα από τη Σύνοδο Κορυφή αυτή. Αλλά τι άλλο έδειξε το Σαββατοκύριακο. Τα κράτη-μέλη βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστικά ως ένα ATM. Όσο γίνεται λιγότερα να καταθέτουν και όσο γίνεται περισσότερα να ε, ε, τραβάνε για όλα τα κράτη-μέλη. Οι φιδωλοί θέλουν να πληρώνουν όσο γίνεται λιγότερα, οι άλλοι να παίρνουν όσο γίνεται περισσότερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι μηχάνημα αυτόματης ανάληψης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είναι ε, μια ένωση που να εγγυάται το μέλλον. Ε, Εράσμους, ε, παιδεία, έρευνα, γνήσια ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι αυτό του υδρογόνου. Θα πρέπει να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που είναι ασθενή τα κράτη-μέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, όμως υπάρχει ένα κράτος μέλος που θέλει να πλουτίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν υπάρχει ένα τέτοιο κράτος μέλος, πρέπει εμείς να έχουμε ένα μηχανισμό διάσωσης, έτσι ώστε τα χρήματα να μην πηγαίνουν σε ε, διεφθαρμένους φίλους κάποιων επίδοξων ε, αυτοκρατόρων. Μέρκελ και Σία ε, γονάτισαν μπροστά στον Όρμπαν σε αυτή τη σύνδοκορυφή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπέκ. Ε, πρώτα τα καλά νέα. Το Brexit έσωσε τη Βρετανία από 80 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά, περίπου όσο θα κόστιζε το Ταμείο για τη Βρετανία. Μην αφήνεις ποτέ μια καλή κρίση να πάει χαμένη. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2027 δαπανά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 750 χρέη. Ε, αυτό είναι πραγματικά πραξικόπημα. Τι λένε τα άρθρα 3.10 και 3.11 τη της για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως και προπολογισμό για την Ένωση αποκλειστικά από ιδίου πόρου. Σαφήνεια. Παράνομα όμω, ε, πάει σε δανεισμό η Ένωση. Ο Κομφούκιο λέει όπου τα λόγια χάνουν το νόημά τους, ε, χάνουν οι λαοί την ελευθερία τους. Όχι στην Ουγγαρία και την Πολωνία, αλλά μέσω των Βρυξελών και του Βερολίνου. Η Μέρκελ συμπεριφέρεται, λες και η Γερμανία είναι πανί ισχυρή, παντοδύναμη όπως οι ΗΠΑ μετά τον πόλεμο και ε, μοιράζει και επιβάλλει ε, ε, φόρους στη Γερμανία για να τα πάρουν άλλοι. Οι Γερμανοί έχουν τη μικρότερη ιδιωτική περιουσία της Ευρωζώνης, τους ψηλότερους φόρους του κόσμου, ε, ηλεκτρικό ρεύμα που κοστίζει στη μέση ρεκόρ και το πιο χαμηλό δίκτυ ιδιοκατοίκησης και ιδιοκτησίας. Ε, η Γερμανία, η πλούσια Γερμανία έχει φτωχούς πολίτες. Ε, τρεις γυναίκες κυβερνάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά είναι πιο ακριβές τρεις γυναίκες από την εποχή της κυρία Μαντάμ του Η κυρία Ντεσούτερ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε Φοντερ κύριε Πρόεδρε Μισε. Ναι, είναι ιστορική η συμφωνία φυσικά και το αναγνωρίζουμε. Αλλά επειδή είμαι γιατρό, πρέπει να πω ότι έχω απογοητευτεί ω γιατρό για τι περικοπέ στο πρόγραμμα τη υγεία. Είμαστε στη μέση τη κρίση, μάλιστα στην αρχή του δευτέρου κύματο. Βλέπουμε όλοι να αυξάνονται τα κρούσματα. Αυτό δεν μπορώ ούτε να το καταλάβω, ούτε να το εξηγήσω στου συναδέλφου μου, γιατί τα κράτη-μέλη δεν το θεωρούν απόλυτη προτεραιότητα. Και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε του αριθμού στην σημερινή πρόταση με προηγούμενα αριθμού αριθμητικά στοιχεία, γιατί δεν είχαμε τότε COVID. Είμαι καθηγήτρια και ερευνήτρια και δεν μπορώ να εξηγήσω στου φοιτητέ μου γιατί έχουν γίνει περικοπέ στο Εράσμο. Δεν μπορώ να εξηγήσω στου συναδέλφου μου ερευνητέ γιατί το Horizon EU δεν είναι αυτό που θα έπρεπε. Γιατί το χρειαζόμαστε για τις καινοτομίε, τι νεοφυεί ε, επιχειρήσεις, τι μικρομεσαίες, να είμαστε ηγετική δύναμη στον κόσμο. Εάν ε, πιστεύαμε την φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή μετάβαση, για την Πράσινη Συμφωνία. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που είναι στραμμένες προς το μέλλον και μας λείπουν από την πρόταση αυτή. Σας παρακαλώ, αν διαπραγματευτούμε το πολιετές και εσείς, ακούστε μας και αυξήστε αυτά τα ουσιαστικότατα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Έπινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, τελείωσε με τα ε, προδοσία του κυρίου Ρούτε. Μετά από διάφορες και αμαχίες τεσσάρων ημερών γονάτισε και γύρισε πίσω. Ε, παρά τους Βρετανούς έχουμε τώρα το μεγαλύτερο το προπολογισμό. Ευρωπαϊκούς φόρους, ευρωπαϊκούς όμους ε, που ε, τόσο καιρό διαρριγνύει τα μάτια του ο κύριος Ρούτε. Είναι φάρσα αυτή η διαδικασία με το φρένο. Μεταφορά πιστώσεων, μεταβιβάσεις, αυτή είναι η Ένωση. Η Ισπανία βάζει κατώτατο εισόδημα, η Γαλλία κάνει άλλες κινήσεις και μειώνονται οι Ολλανδικές συντάξεις. Αυτό είναι πικρό για αυτούς τους ανθρώπους και δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό ζητώ ένα δημοψήφισμα στην Ολλανδία για αυτό το ε, ταμείο και το σχέδιο αναδιανομής του πλούτου να αποφασίζει ο κόσμος μόνος του για τα λεφτά του. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Ντέιλι. Ντέιλι, για ένα λεπτό. Όπως ε, ξέρετε, χτες ε, ο γιατρός Σαΐντ πέθανε στο Δουβλίνο 60 ετών, ένα από τα πολλά θύματα αυτής της υγειονομικής κρίσης και οφείλω να πω πως ε, με συγκλονίζει η απουσία κάθε επαφής ε, μεταξύ των όσων λέτε και της πραγματικότητας για τους πολίτες ε, της Ευρώπης περάσαμε και περνάμε ακόμα μια υγειονομική κρίση άνευ προηγουμένου. Η Κομισιόν μας είπε ότι χρειαζόμαστε το Μάιο 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ για ένα υγειονομικό πρόγραμμα. Η πρώτη δόση των 70 δισεκατομμύριων ανταυτού τίποτα για την υγεία και 1,7 δισεκατομμύρια μόλις στο ΠΔΠ, ενώ 13,5 δισεκατομμύρια πηγαίνουν στην αμυντική βιομηχανία. Τι προσβολή αυτή στον γιατρό που πέθανε. Μιλάτε για αλληλεγγύη, αλλά οι όροι τους οποίους θέτετε εμένα μου θυμίζουν λιτότητα. Λυπούμε, αλλά πρόκειται για μνημείο υποκρισίας. Για 1,5 λεπτό η κυρία Πονσάτη Ομπιόλς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η συμφωνία στο Συμβούλιο Ευρωπαίοι. Οι πολίτες χρειάζονται το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να αντιμετωπίσουν το μέλλον με αισιοδοξία. Αλλά για να επανεκκινήσουν οι οικονομίες μας ε, χρειάζεται κάτι περισσότερο από σκληρή δουλειά και χρήματα. Πρέπει να προωθήσουμε το δυναμικό, το δημιουργικό που έχουμε. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία και την επιστήμη. Και όμως έγινε το αντίθετο περιεκόπιο ο προπολογισμό της έρευνας. 27 πρωθυπουργοί δεν το συνειδητοποίησαν. Ζητάω λοιπόν από το Κοινοβούλιο να υπεραστεί τον προπολογισμό της έρευνας ε, και το κράτος δικαίου εγκαταλειφθήκε αλλά χαίρομαι για το ότι τουλάχιστον εγκρίθηκε ένας μηχανισμός ελέγχου. Η Ισπανία θα λάβει πολλά χρήματα, χρήματα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά. Και ναι, απαιτείται εξωτερικός έλεγχος, γιατί η Ισπανία είναι το κράτος μέλος όπου ο βασιλικός οίκος είναι το επίκεντρο ενός σκανδάλου διαφθοράς το οποίο αρνείται το Κοινοβούλιο να διερευνήσει ξοδεύει δισεκατομμύρια σε υποβρύχια που δεν μπορούν να δέσουν στο μόλο και αεροπλάνα που δεν πετάνε. Φτιάχνει τρένα υψηλής ταχύτητας ενώ οι τοπικές συγκοινωνίες δεν λειτουργούν. Είναι η χώρα η οποία διασώζει τις τράπεζες και όχι τον λαό. Χαίρομαι λοιπόν που κάποιος θα κοιτάει και θα παρακολουθεί πώς θα ξοδευτούν αυτά τα λεφτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χαλίτσκι για δύο λεπτά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια και σε εσά κυρία Πρόεδρε, γιατί η Σύνοδος Κορυφής ε, στέφθηκε με επιτυχία. Είναι μια ιστορική στιγμή που τόσο δαψιλά κονδύλια, δυνητικά, αλλά ελπίζω τελικά να πραγματοποιηθούν, ε, θα μπορέσουν να διασώσουν την ευρωπαϊκή οικονομία για να ανακάμψει μετά την κρίση του κορονοϊού. Πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα προστατευτούν και από τον μηχανισμό του κράτου δικαίου. Αυτό είναι επιτυχία. Αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τον πολιετή προπολογισμό, το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, που στόχο έχει να υλοποιήσει του στόχου μα. Πώς είναι δυνατόν όμως ε, με το ένα χέρι να υπογράφουμε περικοπές στο Ταμείο Δικής Μετάβασης που κανονικά θα χρησιμεύσει για να υλοποιήσουμε το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Και να λέμε ότι είναι προτεραιότητά μας αυτό, οι περιφέρειες που εξαρτώνται από τον άνθρακα, όπως η Σιλισία, ε, θα πρέπει τέτοια ταμεία, όπως το Ταμείο Δικής Μετάβασης, να το ενισχύουμε, όχι να το αποδυναμώνουμε. Δεν μπορούμε να λέμε στους νέους συμπολίτε μας ότι η Ευρώπη τους σκέφτεται, φροντίζει για την παιδεία τους και ταυτόχρονα να περικόπτουμε κατά 60% το πρόγραμμα Έρασμος που είναι το ευληματική πρωτοβουλία της ε, σύγχρονης, ανοιχτής, ε, ε, καινοτόμου Ευρώπης που επενδύει στην παιδεία. Επίσης, ε, έχουμε ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου που σκοτώνει περισσότερο ε, στην Ευρώπη από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Και με τον κορονοϊό είχαμε μεγάλες υγειονομικέ προκλήσεις. Αλλά ουσιαστικά ακυρώσαμε την οικονομική μας πολιτική στο νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνήσει σε αυτό. Πολλά λέμε για το κράτος δικαίου. Και αν είναι τόσο σημαντικό το κράτος δικαίου και αν κοπτόμαστε για το κράτος δικαίου, ε, το πρόγραμμα δικαιώματα και αξίες που προωθεί τη δημοκρατία και τις ε, θεμελιώδεις αξίες θα πρέπει να ενισχυθεί όχι να αποδυναμωθεί. Έχουμε την ε, προστασία των εξωτερικών συνόρων και άλλα θέματα. Ε, θέλουμε αλληλεγγύη στην Ευρώπη, αλλά να μην ξεχνούμε τι προτεραιότητε και τη χρηματοδότησή του, Γι' αυτό θα πρέπει να διορθώσουμε τον πολίτη προπολογισμό. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Γκαρδιασάμπαλ Ρουμπιάλ. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε Φοντερ Λάιεν, κυρία Πρόεδρε Μισελ. Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια συνήθως δημιουργούν πολλές προσδοκίες και πολλές φορές και απογοητεύσεις και ε, ματέωση, κάτι που δεν ίσχυσε όμω την τελευταία φορά. Μπράβο σα, συγχαρητήρια ήταν καταπληκτικό το έργο σα. Καταλήξατε σε ιστορική συμφωνία και επιτέλου ε, είχατε το κουράγιο να κάνετε αυτό που έπρεπε. Κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Κάτι που περιποιεί τιμή σε αυτή τη φράση του Μονέ, που λέει ότι η Ευρώπη χτίζεται και οικοδομείται στι κρίσει. Το σχέδιο ανάκαμψη είναι μικρότερο από ό,τι περιμέναμε και το Ταμείο. Ε, είναι σημαντικό παρόλα αυτά και ελπίζω να είναι και επαρκέ. Αυτό που είναι ανεπαρκέ είναι το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί κάνατε λάθο. Δεν μπορεί για τρίτη φορά να έχουμε προπολογισμού ε, ε, μικρότερου από την προηγούμενη επταετία. Ενώ οι ανάγκε μα είναι όλο και μεγαλύτερε. Και εδώ δεν μιλώ για τι ανάγκε που δημιούργησε η κρίση του κορονοϊού, γιατί γι' αυτό έχουμε το σχέδιο ανάκαμψη. Πριν το κορονοϊό όμω επίση είχαμε πολλέ ανάγκε και θα πρέπει και αυτέ να τι χρηματοδοτήσουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε την έρευνα για το Αλτσχάιμερ, για τον καρκίνο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε καινοτόμα βιομηχανικά σχέδια, πιο αποτελεσματικά μέσα μεταφορά και τρόπου μεταφορά. Να δώσουμε κατάρτιση στου ανέργου, να βοηθήσουμε του νέου να εισέλθουν στην αγορά εργασία, να καταπολεμήσουμε την παιδική φτώχεια. Αυτέ είναι ανάγκε που υπάρχουν ακόμη και γι' αυτό χρειαζόμαστε στιβαρού προπολογισμού. Και είναι κρίμα που αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα που διείπε την Ευρωπαϊκή, το, την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής υπέκυψε τελικά σε αυτή την αμήλικτη λογιστική. Ελπίζω τελικά να καταλήξουμε σε συμφωνία και πραγματικά ελπίζω να είναι ουσιαστικά και τέλεια στο προπολογισμό. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριο Σφερχόφστατ για 1,5 λεπτό. Πρέπει να σας πω ότι κάποτε ήμασταν κάτι μοναχικοί καβαλάριδες που από την αρχή της κρίσης ε, του ευρώ ότι χρειαζόμασταν ευρωομόλογα και νέους ιδίους πόρους και όλοι έλεγαν είστε ονειροπόλοι, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό, αυτή είναι η Ευρώπη, τι είναι αυτά που λέτε, ε, ανεδαφικά, είστε φεροβάμονες. Μα ορίστε, έγινε πραγματικότητα και είναι ιστορική. Το, πρώτο άλμα ήταν η ενιαγορά, αγορά, η δεύτερη το ευρώ και το τρίτο είναι ότι εκδίδει για πρώτη φορά ομόλογα η Ευρώπη και θα αυξήσει την δημοσιονομική της δυνατότητα ε, με τρόπο πραγματικά δραματικό και, τεράστιο. Υπάρχουν και αδυναμίες προφανώς και η μεγαλύτερη αδυναμία οφείλεται στον κανόνα της ομοφωνίας. Γι' αυτό το λόγο τα πανευρωπαϊκά προγράμματα έχουν περικοπεί και έχουν αυξηθεί οι άμεσες μεταβιβάσεις και παραμένουν επιστροφές για τους φιδωλούς. Θα είμαι εδώ πάρα πολύ ομός αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματος όλου του Κοινοβουλίου. Εγώ δεν βλέπω τούτο εδώ το Κοινοβούλιο να δίνει πράσινο φω για το πακέτο αυτό και για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αν δεν διορθωθεί. Ε, και πάλι τα πανευρωπαϊκά προγράμματα αν δεν γίνουν και πάλι προτεραιότητα στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και είναι εύκολο να γίνει. Ποιο είναι το εύκολο, να αρχίσουν νωρίτερα οι ήδη πόροι από ό,τι προβλέπεται στο σχέδιο. Το σχέδιο λέει το 2023. Προτείνω να αρχίσουν από το 2021. Και τέλος, πρόεδρε, πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι ε, το όπλο σας και το σφυρί σας εναντίον μου όπως κάνετε κάθε φορά είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει συναπόφαση με το κοινοβούλιο. 750 ε, δισεκατομμύρια θα δαπανίσουμε και θα συλλέξουμε. Αυτό γίνεται μόνο με δημοκρατικό έλεγχο. Στην Ευρώπη είμαστε, ούτε στη Ρωσία ούτε στην Κίνα. Thank you. It was good... Ευχαριστώ. Ε, μπράβο κύριε Φερχόφστατ και δεν σας έκοψα, διέκοψα κιόλα. Εντάξει, ε, κοντεύουν διακοπές. Ε, λεπτό ο κύριος Μάγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζούμε σε ιδιαίτερου καιρού. Νομίζω αυτό το ξέρουμε όλοι. Και ιδιαίτεροι καιροί χρειάζονται φυσικά και ιδιαίτερα μέτρα. Εδώ πρόκειται για πολλά. Ε, Δηλαδή έχουμε το 1 με 12 μηδενικά. Ε, πολλά διακυβεύονται εδώ. Αυτά τα πακέτα και αυτές οι αποφάσεις θα καθορίσουν και θα επηρεάσουν ε, την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική γενεών μετά από μας. Και κατά περίεργο τρόπο όλοι βγαίνουν νικητές από αυτό. Μέρκελ, Κούρτς, Μακρόν γύρισαν στις πρωτεύουσές τους και δήλωσαν ότι κέρδισαν στις διαπραγματεύσεις για τις χώρες τους. Κάτι πέτυχαν. Βέβαια όποιος έχει διαπραγματευτική και το λέει και η κοινή λογική ε, αυτό δεν μπορεί να, να εμφανίζεται ως νικητής οι πάντες. Η Γαλλία και η Γερμανία λέει σε τελική ανάλυση κερδίζουν από αυτά τα μέτρα γιατί έχουν αλλάξει τα κριτήρια ε, ε, με βάση το μέγεθος και μας απορεί πραγματικά μας προκαλεί έκπληξη, έκπληξη συγγνώμη, ότι όλοι εμφανίζονται ως νικητές. Και από αυτές τις τσέπες, τις πολλές και μεγάλες τσέπες, τι έχουμε τώρα, μια ένωση χρεών. Αυτή συνάδει με τις συνθήκες. Χρειάζεται να ελεγχθεί. Το είπαν αυτό, το επενήχθησαν κάποιοι συνάδελφοι. Γιατί το κράτος δικαίου δεν μπορεί να ισχύει μόνο για τους άλλους, θα πρέπει να ισχύει και για τους εαυτούς μας, αγαπητοί συνάδελφοι. Αξιότιμοι. Πάντως, τι ε, είναι ξεκάθαρο, ότι δημιουργούμε τώρα ένα, ε, διάφορα μπλοκ, βορράς, νότος, ανατολή, δύση και υποτιθέμενη ένωση αλληλεγγύης που θέλετε, ε, ε, αυτό είναι ε, μειονέκτημα. Η αλληλεγγύη ποτέ δεν μπορεί να είναι μονόδρομος, αξιότιμη συνάδελφοι. Για ένα λεπτό η κυρία Χάν. Είναι θετικό το ότι έχουμε τώρα μια διαπραγματευτική θέση και είναι ένα ισχυρό μήνυμα για το ότι θα στηρίξουμε την Ευρώπη. Αλλά οι διαπραγματεύσεις τώρα ξεκινάνε. Δεν είναι αποδεκτό να έχουμε περικοπές σε αυτά τα οποία αφορούν το μέλλον στην υγεία και στην έρευνα και να μην υπάρχουν όροι για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου και πολύ λίγα λεφτά για το κλίμα. Πρέπει να σώσουμε την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη το αργότερο μέχρι το 2050 με ένα Green Deal για να επανεκκινήσει η οικονομία. Να σταματήσει η βιομηχανία να εκπέμπει άνθρακα. Χρειάζεται λοιπόν έρευνα γι' αυτό. Να στηρίξουμε τις μικρές και μεσαίες ε, επιχειρήσεις. Ε, δεν μπορούμε πλέον να έχουμε ορυκτά καύσιμα. Ο πρόγραμμα ορίζοντας. Όλα αυτά είναι μέσα για το μέλλον. Έχουμε υποσχεθεί ότι θα σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων με ένα ισχυρό ταμείο για μια δίκαιη μετάβαση. Κάποιε περιφέρειε ήδη κάνουν κάποια σχέδια μετάβασης και το Συμβούλιο τους αφήνει ξεκρέμαστους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να γίνει το μεγάλο βήμα προς μια αλληλέγγυα η οικονομία με όλες τις θετικές ευκαιρίες που αυτό σημαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λούντγκρεν για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι το πακέτο η δέσμη μέτρα του Συμβουλίου αντιβαίνει στο άρθρο 311 της Συνθήκης. Εκεί αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δανειστεί χρήματα για να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό της και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει για την τήρηση των κανόνων και να μην αγνοούμε και να ψηφούμε κανόνες και διατάξεις της ίδιας της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μία κατάσταση στη Σουηδία όπου κόσμος πεθαίνει και ταυτόχρονα η Πρωθυπουργός στέλνει χρήματα στο εξωτερικό με 6 δισεκατομμύρια που θα συμπληρώσουμε στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό είναι επιστροφή. Και τώρα μιλούμε για φορολογία και ίδιους πόρους. Ξεπουλήσατε τη Σουηδία και τους Σουηδούς. Ελπίζω να λάβουν υπόψη αυτό οι ψηφοφόροι Ο κύριος Μποτανγκά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Φόντερ Λάιν, κύριε Μισελ. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα δανειστεί από κοινού για να τα βάλουμε όλα ε, σε ένα ταμείο και με τα βιβάσεις να πηγαίνουν στις χώρες που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και απέναντι στους διαφόρους Μαρκ Ρούτε του κόσμου τούτου που δεν θέλουν να δείξουν την παραμικρή αλληλεγγύη σε αυτή την πανδημία. και το μόνο που κοιτάνε ε, είναι πότε φεύγει κανείς στη σύνταξη και ε, σε ποια ηλικία σύνταξη δοτείται. Ε, όμως θέλω να σας προειδοποιήσω γιατί το βάλετε αυτό στο ευρωπαϊκό εξάμεινο αυτή την ελάχιστη ελεγγύη. 63 φορές τα κράτη-μέλη έχετε δώσει συμβουλές και συστάσεις να περικόψουν τους προϋπολογισμούς για την υγεία. Αν ε, προχωρήσετε ακόμα αυτά τα ανταλαϊκά, αντιλαϊκά και αντικοινωνικά μέτρα θα μας βρείτε απέναντί σας όταν στρέφεστε κατά των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ. Thank you. One minute, Mr. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Καστάλντο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο μαραθώνιος του Συμβουλίου τελείωσε με μια συμφωνία η οποία ε, θέλει να αντιμετωπίσει με δύναμη και αποφασιστικότητα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Έχουμε όμως ε, το πρόγραμμα αυτό το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα λάθη της ε, λιτότητας και θα θέλαμε εδώ πέρα να επενέσουμε τον πρόεδρο Κόντε για τα όσα έκανε απέναντι στις φιδωλές ε, χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να μην οδηγηθούμε και πάλι σε ένα χρονιστικό όργανο διακυβερνητικό. Τα προγράμματα για την Ευρώπη, το αύριο, το Horizon Europe, EU for Health, Erasmus Plus λοιπά. δεν θα έπρεπε να έχουν περικοπή. Και βεβαίως ε, βλέπουμε ότι θα πρέπει να επιβληθεί φόρος ε, άνθρακα στα σύνορα. Δεν πρέπει να διστάζουν οι ηγέτες μας. Ως κοινοβούλιο εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την μάχη. Γι' αυτό λοιπόν η διάσκεψη αυτή για το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να φέρει μία αναθεώρηση των συνθήκων. Γιατί όσο υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο δεν θα μπορέσει ποτέ να νικήσει η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Σάιερ. Ε, με μικρόφωνο παρακαλώ. Σας ε, ευχαριστώ. Ε, πάρα πολλοί μιλάνε εδώ πέρα για κράτος δικαίου. Ε, δεν ξέρω εάν ε, ξέρουν τι σημαίνει η λέξη. Κράτος δικαίου σημαίνει ελευθερία και δημοκρατία και το να ε, υπερισχύει το δίκαιο. Η γενιά μου πριν από 30 χρόνια πάλεψε γι' αυτό έτσι ώστε να μην είναι κάτι τέτοιο προνόμιο της Δυτικής Ευρώπης. Πολεμήσαμε γι' αυτό, αλλά πρέπει να σας πω τι δεν σημαίνει κράτος δικαίου. Αυτό για το οποίο θέλετε να το χρησιμοποιήσετε εδώ πέρα. Να επικαλείστε κανόνες που δεν είναι γραμμένοι πουθενά. Να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για το ίδιο πράγμα, άλλους να επενούμε και άλλους να κατηγορούμε, δηλαδή να τιμωρούμε την ιδεολογία. Αυτό θέλουν κάποιοι να κάνουν και να τα υποτάξουν όλα αυτά σε κομματικά κριτήρια. Αν είναι έτσι, δεν μπορεί να αλλάζουμε τους κανόνες της ε, ψηφοφορίας για να δημιουργούμε κάτι το οποίο θέλουμε να επιτυχούμε όπως έγινε στην ε, έκθεση Σαρτζεντίνη. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την αντίθετη γνώμη και ο κατηγορούμενος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αντιδράσει και να υπερασπιστεί αυτόν. Ε, αρνηθήκατε να απαντήσει ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Νούλα πένα σύνε λέγε. Δεν υπάρχει τιμωρία χωρίς νόμο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτό. Δεν υπάρχουν νομικά κριτήρια. στην, περίπτωση μιας υποψίας ε, θα επιληθούν κυρώσεις και δεν υπάρχει ίση μεταχείριση. Αυτό είναι κομμουνιστικό μοντέλο. Είναι μια αστυνομία σκέψης όπου τιμωρείται η πρόθεση. Αυτό είναι σοβιετική μέθοδος κατάχρησης του νόμου για εκβιασμό. Το ξέρουμε, τα αναγνωρίζουμε, έχουμε ήδη υπάρξει θύματα αυτής της ε, μεθόδου, το νικήσαμε και δεν θα επιτρέψουμε να ξαναέρθει από την πίσω πόρτα. Η Ευρώπη αξίζει κράτος δικαίου. Εδώ πέρα κάποιοι πολιτικοί λένε ψέματα για το ότι τηρούν τους κανόνες στο όνομα του κράτους δικαίου. Όμως το κοινοβούλιο αυτό παραβιάζει τους κανόνες τους και τον κανονισμό του, τα άρθρα 132 και 127 που λένε σαφώς ότι η ψηφοφορία μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν τελειώσει η συζήτηση. Εμείς συζητάμε ακόμα και έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Έχουμε παραβίαση του κανονισμού εδώ, των αξιών μας. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε πρώτα τα του οίκου μας και μετά κάνουμε μαθήματα στους άλλους. Σας ευχαριστώ κύριε Σάιρ η τελική ε, ψηφοφορία θα γίνει μετά την συζήτηση, λέει η πρόεδρος. Περνάμε τώρα στον κύριο Φερνάντες για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των τελευταίων ημερών συνιστά ένα ιστορικό βήμα υπερβατικού χαρακτήρα στην πορεία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Μία συμφωνία που ουσιαστικά είναι η συνέχεια στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο ψήφισμα του Μαΐου. Εκεί απαιτήσαμε την δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού μέσω κοινοτικού δανεισμού και ε, χρηματοδότηση με ιδίους πόρους για να αντιμετωπίσουμε την κρίση σημαντική πρόταση θεμελιώδης σημασία που η κυβέρνηση τη Ισπανία ε, υπό την ηγεσία του Πέντρο Σάντσες διαδραμάτισε κέριο ρόλο. Έχουμε όμως κάποια θέματα αμφισβητούμενα. Το πρώτο είναι ο τακτικός προπολογισμό. Μερικά τμήματα δεν αυξάνονται όπως θα έπρεπε. Ιδιαίτερα το Ταμείο της δίκής Μετάβασης, όπου οι χώρες ε, και οι περιφέρειες όπως η Αστούρια, ε, η γενέτειρά μου, που θέλουν να, να εξυγχρονίσουν την οικονομία του και θα πρέπει να κάνουν τεράστιε προσπάθειες, θα πρέπει να στηριχθούν αντίστοιχα. Επίσης, ε, ο μηχανισμό ανάκαμψη ε, και ανθεκτικότητα, που θα βοηθήσει τις χώρες στην πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων έχει μια διακυβέρνηση ε, μόνο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι που δεν δέχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε διακυβέρνηση με σαφή δημοκρατική νομιμοποίηση, όπου θα εκπροσωπούνται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και εκεί θα έχει το λόγο του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα βρεθούμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στου τριμερεί διαλόγου πριν το τέλο του έτου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για 1,5 λεπτό, ο Σεζορνέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία φυσικά είναι ιστορική, το είπαν όλοι. Μπορεί να διαφωνεί η ακραδεξιά. Ο, κύριε Μπέ, σίγουρα μπορεί να μην είναι δική σας ιστορία, αλλά είναι δική μας. Και σίγουρα αντικατοπτρίζει η συμφωνία αυτή την εξαιρετική όθηση ε, και μια, ένα σχέδιο ανά, ανάκαμψης μαζί με τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Μην ξεχνάτε από πού ξεκινήσαμε. Πριν από λίγε εβδομάδε μα έλεγαν ότι είναι ανέφικτη συμφωνία, αποκλείεται. Μερικοί έβαλαν βέτο ακόμη και επί τη αρχή ενό έκτακτου σχεδίου ανάκαμψη ε, κατά των ε, μεταφορών, κατά την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ε, ανάληψης χρέους και τελικά τα καταφέραμε, κάτι που είναι άξιο συγχαρητηρίων και αξιοθαύμαστο. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το λεπτό καθήκον να χαιρετήσει αυτή την ιστορική συμφωνία, υπενθυμίζοντα όμω τα αιτήματα των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών λαών. Γιατί αυτό είμαστε εμεί οι Ευρωβουλευτέ. Είμαστε θετικοί απέναντι στη συμφωνία. Ταυτόχρονα όμω είμαστε και η 28η φωνή σε αυτέ τι διαπραγματεύσει, σε αυτή τη συζήτηση. Και θα προτείνουμε ε, εύλογε τροποποιήσει ε, συγκεκριμένε, περισσότερα κονδύλια για το έρασμο, περισσότερα κονδύλια για την υγεία και κυρίω περισσότερου ιδίου πόρου αποτελεσματικού και πιο γρήγορα. Και συμφωνώ με τον ε, συνάδελφο Κίφερ Χόφστατ. Πιο γρήγορα θέλουμε ιδίου πόρου για να αποπληρώσουμε το κοινό μα χρέο. Ακούσαμε ότι τέσσερι μέρε συζήτηση μεταξύ των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων ήταν το τίμημα τη δημοκρατία. Συμφωνώ. Πουθενά σε άλλη ήπειρο 27 χώρε ε, μέλη κατάφεραν να συμφωνήσουμε σε τέσσερι μέρε για τόσο φιλόδοξο σχέδιο. Έχουμε όμω μπροστά μα κάποιε εβδομάδε διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έναν προπολογισμό που θα, μα δεσμεύσει για μια επταετία. Και αυτό είναι το τίμημα τη δημοκρατία. Δεν θα μπλοκάρουμε τον προπολογισμό, αλλά θα δηλώσουμε παρόν στο ραντεβού τη ιστορία. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριο Βαντεντρίσε. Πρόεδρε, συνάδελφοι, 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά ε, θα πρέπει να δώσει καθαρά το Βέλγιο για το Ταμείο Ανάκαμψης από τον κορονοϊό. Επίσης αυξάνεται κατά ένα δις και πλέον ετησίως ε, η συμμετοχή μας. 50 δις ε, περικοπές και 130% δημόσιο χρέος έχουμε. Αυτό πώς να το εξηγήσω στους πολίτες, στους ψηφοφόρους μου, ότι δεν έχουν χρήματα για τις συντάξεις, για την υγεία, για δέκα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που κινδυνεύουν, αλλά υπάρχουν δισεκατομμύρια για την πολιτική του Άι Βασίλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ούτε εσείς ή μήπως περισσότερο. Όσο περισσότερη εξουσία έχουν οι ευρωκράτες επί των κρατών, τόσο καλύτερα μπορείτε να ελέγχετε τα πράγματα. Ε, δημιουργείται εξάρτηση από κάποιους που δεν έχουν ε, ποτέ εκλεγεί. Αυτοί οι ευρωφανατικοί ε, χάνουν δημοψηφίσματα, σαμποτάρουν, εκβιάζουν για τον Brexit. Τίποτα δεν πιάνει. Ποια είναι η δημοκρατία και η ελευθερία. Τώρα ευρωπαϊκό χρέος και ευρωπαϊκούς φόρους θέλετε να εισάγετε. Με αυτόν τον τρόπο ε, θέλετε να χρηματοδοτήσετε και να γίνει μια φυλακή η Ευρώπη, φορολογική και δημοσιονομική. Και κανείς δεν θα μπορεί να ξεφύγει. Για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς ποτέ δεν θα ψηφίζαμε. Ε, για ένα λεπτό η κυρία Μέτς. Αξιότιμη πρόεδρη, Κυρία Πρόεδρε, εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχει σαφής πλειοψηφία για περισσότερη ελεγγύη, για περισσότερη διαφάνεια, για περισσότερη βιωσιμότητα, για περισσότερη Ευρώπη. Το θέμα δεν είναι ποια χώρα θα πάρει πόσα και γιατί και τι. Το ερώτημα είναι σε τι θα επενδύσουμε. Η διάσωση της οικονομίας δεν μπορεί να είναι εις βάρος κάποιων προγραμμάτων του μέλλοντος. Πώς μπορούμε να μιλάμε για την επόμενη γενιά και μειώνουμε τις δαπάνες στην παιδεία. Πώς θα εφαρμόσουμε μια πράσινη συμφωνία ε, αν ε, μειώνουμε στο μισό τον προϋπολογισμό ε, το σχετικό για τη δίκαιη μετάβαση. Πώς μειώνουμε τα κονδύλια για την υγεία και για την έρευνα και τα διαγράφουμε. Τι γίνεται με τις ελπίδες μας για μια κοινή γεωργική πολιτική πιο βιώσιμη όταν μειώνεται στο μισό ε, η στήριξη του δεύτερου πυλώνα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να τα υποστηρίξει ως περίκοπες. Γιατί όταν έχουμε ενοικοδόμηση, κατά τη διάρκεια της γίνεται ακριβώς η ενοικοδόμηση, όχι μετά από αυτήν. Ε, για ένα λεπτό, κύριο Φιντάντσα. Σας ευχαριστώ. Φιντάντσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από την ρητορική και την ε, θριαμβολογία χρειάστηκαν λίγες ώρες για να ανακαλύψουμε ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία αυτή. Τα ε, βλέπετε εδώ πέρα. Βεβαίω, ε, εντάξει, χθε είχαμε κάποια χειροκροτήματα, Χειροκροτούσα χθε ο τον κύριο Κόντε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Αλλά βλέπουμε ότι είναι λάθο να συνεχίζουμε με τι εθνικέ ε, εκπτώσει, πω θα φτάσουν πάρα πολύ αργά τα λεφτά όταν θα έχουν κλείσει ήδη πάρα πολλέ επιχειρήσει και χρειάζεται ένα μηχανισμό για να βοηθήσουμε άμεσα. Πρέπει λοιπόν να καταγγείλουμε την διακυβέρνηση η οποία θέτει εν κινδύνο την οικονομική μας ε, πολιτική και πάλι βεβαίως ε, μένουν ε, χωρίς ανταγωνισμό οι Κινέζοι και οι τεράστιοι οικονομική όμιλοι. Και τι έχουμε τελικά, ένα φόρο στα πλαστικά. Αυτά ε, τα έχετε γράψει εσείς, όχι εγώ. Σας ευχαριστώ, Εστάρα Σαραγκούτη για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να στείλω τη στοργή μου και την υποστήριξή μου στις οικογένειες των θυμάτων το κρατούμε στη μνήμη μα. και επίση να αποτίσω φόρο τιμή ε, στου εργαζόμενου ε, που έδιναν και δίνουν τη μάχη του κατά τη πανδημία. Είναι θετική η συμφωνία, κάνει βήμα προόδου και δεν θα πρέπει να χάσουμε ούτε ένα λεπτό γιατί ο χρόνο μα πιέζει και ήδη έχουμε καθυστέρηση. Θα πρέπει λοιπόν με θάρρο και ταχύτητα να δράσουμε. Πρόκειται για ένα σχέδιο ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αλλά και ευρωπαϊκή συνοχή. Είναι και μια ιστορική συμφωνία γιατί ουδέποτε στο παρελθόν είχαμε μια τέτοια κοινή συμφωνία των κρατών μελών και έχει και τεράστιε διαστάσει ε, και τα κονδύλια. Σαφέστατο στόχο. Ανάκαμψη τη της επασχόληση. Προστασία τη Ευρώπη ε, των ζώων. Ανάκαμψη. Χάρη στην, στον ηγετικό ρόλο της καγκελαρίου Μέρκελ και της ε, ε, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι δύο γυναίκες και μάλιστα του Λαϊκού Κόμματο. Έχουμε λοιπόν ένα φιλόδοξο και στιβαρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να δείξουμε αυτή τη φιλοδοξία. Στο παρελθόν το κάναμε στην Ισπανία με το Ραχώη. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε την ευθύνη τη και έκανε το καθήκον του. Τώρα θα πρέπει το ίδιο να κάνουν και τα κράτη-μέλη απέναντι στου πολίτε. Κυρίω η Ισπανία θα πρέπει να πριτανεύσει το γενικό συμφέρον και να αφήσουμε του αγώνε ε, ε, ή τι ισορροπίε τη εξουσία. Και επίση τα κονδύλια να δαπανηθούν εκεί που χρειάζονται. Τώρα, το δεύτερο τμήμα τη συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο δεν μα ικανοποιεί. Είναι αδικαιολόγητε κάποιε περικοπέ. Το 10% η περικοπή στη γεωργία και στην αγροτική ανάπτυξη είναι αδικαιολόγητη. Δεν μπορεί ε, η αγροτική ανάπτυξη να θυσιαστεί στο βωμό της συμφωνίας, ιδιαίτερα όταν πλήγει στη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης, περικοπές στην υγεία, στην δίκη μετάβαση, στην παιδεία, στο έρασμος, όλες αυτές οι περικοπές διακυβεύουν το μέλλον της Ευρώπης. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι με προβληματίζει ε, πολύ το θέμα της προστασίας του κράτους δικαίου. Θέλουμε μηχανισμούς που θα εξασφαλίζουν την προστασία του κράτους δικαίου. Χωρίς κράτος δικαίου δεν υπάρχει δημοκρατία και χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Πύρη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Επίση, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια θετική χρειά. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα ε, του πρόεδρου Μισελ και Φόντερ Λάιεν για το επίτευγμά του στο σχέδιο ανάκαμψη. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία συμφωνεί ότι το σχέδιο ανάκαμψη είναι καινοτόμο και αυτό χρειάζονται όσοι φοβούνται σήμερα ότι θα χάσουν τη δουλειά του. Συγχαρητήρια λοιπόν για τη διορατικότητα του σχεδίου ανάκαμψη. Αλλά εδώ σταματούν τα εγκομιακοί έπαινοι. γιατί πιστεύω ότι το ΠΔΠ δεν είναι ένα προπολογισμό που ανταπεξέρχεται στο ύψο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Είναι ένα προπολογισμό χωρί φιλοδοξία, χωρί ε, ε, μοντερνισμό δεν είναι σύγχρονο αυτό ο προπολογισμό. Φυσικά και δεν μπορείτε να είστε ικανοποιημένοι, κυρία Φοντερ Λάιεν. Η κρίση αυτή οδήγησε σε παγκόσμια ανισότητα. Και τι κάνουμε, περιορίζουμε τα κονδύλια τη αναπτυξιακή βοήθεια. Και το πιο σημαντικό σημείο, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί για τα χρήματα μπορούμε να διαπραγματευτούμε, αλλά οι αξίε μα είναι διαπραγματεύτε. Και το γενικό ότι έχουμε ηγέτες, καθηγητέ δικαίου, δημοσιογράφου που ερμηνεύουν διαφορετικά τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Αυτό είναι ένα κακό σημάδι. Μερικοί λένε ότι επιτέλους ε, για πρώτη φορά και ευτυχώ αναφέρουμε μαζί τον προπολογισμό και το κράτος δικαίωμα. Δεν έχουμε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Αυτό δεν το χρειαζόμασταν πριν από μία δεκαπενταετία. Σήμερα όμως έχουμε δύο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που με βάση του Freedom House είναι, είναι υβριδικά καθεστώτα και δεν πληρούν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Ελπίζω η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απαιτήσει σαφή διατύπωση για το κράτος δικαίου πριν συμφωνήσει για τον προϋπολογισμό. Και δεν μιλούμε για χρήματα, μιλούμε για αξίες. Σας ευχαριστώ, κυρία Τσέχ, για ένα λεπτό. Ο αρχισυντάκτης, ο ε, του μεγαλύτερου πόρταλ της Ουγγαρίας απολύθηκε χτες ε, λίγες ώρες ε, αφότου ο πρόεδρος Όρμπαν είπε ότι νίκησε τις Βρυξέλλες. Πρόεδρε Μισελ, πρόεδρε Φοντερ Λάιν, κούφια λόγια. Ο προπολογισμό αυτό είναι μια ιστορική ευκαιρία για να ξαναχτίσουμε την Ευρώπη. Και χαίρομαι, αλλά η συμφωνία αυτή θα είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε εμεί. Μπορεί να απειλήσει την Ευρώπη ή τους Ευρωπαίους λαϊκιστές γιατί και χτες δεν υπήρξε κάποιος μηχανισμός κράτους ε, δικαίου που να έχει ξεκάθαρο, ξεκάθαρη σχέση με τον ε, προϋπολογισμό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε άλλα κούφια λόγια, ούτε λεφτά τα οποία θα πηγαίνουν στις τσέπες των ολιγαρχών. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, τα χρειαζόμαστε. Ζητάμε από την Κομισιόν να αναλάβει δράση και ηγεσία επί των ζητημάτων αυτών και ζητάμε από τη Γερμανική Προεδρία να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία υποσχέθηκε η κυρία Μέρκελ και να δει ως πρώτη προτεραιότητα το θέμα του κράτους δικαίου. Οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο για εμάς. Η κυρία Λαπόρτ. Ευχαριστώ κύριε Λαπόρτ. Τέσσερα μερόνυχτα σκληρών διαπραγματεύσεων ε, δεν ένωσαν την Ευρώπη τελικά συμφώνησαν ξυλώνοντας την αρχική πρόταση συμβολική αποτυχία. Αποτυχία για την Ευρώπη με διελκυστίδες και ανταγωνισμούς. Αποτυχία για την αξιοπιστία του εγχειρήματο. Ο Μακρό είπε την Τρίτη το βράδυ ότι υποτίθεται δεν θα πλήρωνε τίποτα ο Γάλλος φορολογούμενος. Ποιος θα πιστεύει αυτά τα παραμύθια με την Ευρωπαϊκή Ένωση περπατάμε πάνω στο νερό. Χρειάζεται ομόφωνη απόφαση για να αναλυφθεί το δάνειο και πώς θα το αποπληρώσουμε. Ε, είναι κατά του άρθρου 310 ε, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαράδεκτα. Φοβάμαι την επόμενη φάση που θα είναι δημιουργία ε, Υπουργείου Οικονομικών στην Ένωση αποτυχία και για τις προτεραιότητες. Πώς θα εξηγήσετε ε, το, ότι μειώνεται το EU for Health που ήταν η απάντηση στην πανδημία. Δεν γνωρίζει σύνορα η πανδημία, κανένα δίδαγμα δεν βγάλαμε. Αποτυχία ως προς τις δεσμεύσεις που δεν δεχόμαστε και δεν τιμούμε. Συνεχίζονται οι επιστροφές. Κανονικά υποτίθεται ότι θα είχαν καταργηθεί. Τελικά θα γίνουν συζητήσεις για την αρχή της επιχωρικότητας. Γιατί ένα ευρωπαϊκό ε, σχέδιο είναι πιο αποτελεσματικό από ε, πολλά εθνικά. Φαίνεται πόσο θνησιγενές είναι αυτό το σχέδιο του φεντεραλισμού για τα έθνη. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος ε, Κόμμα. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ανακουφιστήκαμε γιατί ε, αποτρέψαμε τα χειρότερα, την έλλειψη συμφωνίας δηλαδή που θα επιδίνωνε την κρίση που διανύουμε. Αλλά όπως πολλοί ε, ευρωπαϊστές έχω μια γεύση πικρή, μια γεύση στάχτης στο στόμα γιατί είδαμε εθνικούς εγωισμούς να συγκρούονται. Ε, το συλλογικό ευρωπαϊκό εγχείρημα και θυμικό έχει να βαγίσει, έχει καταρρεύσει. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Σχεδόν δεν υπάρχουν ήδη οι πόροι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δράσει ουσιαστικά. Η διαχείριση του Ταμείου ανάκαμψη πληγώνει την ίδια την ιδέα που έχουμε για τη δημοκρατία. Τελικά λέγει η ε, θυσία των ε, οικολογικών στόχων. Ε, το σχέδιο ανάκαμψης ε, δεν διαφέρει από κάποιο κλασικό σχέδιο. Μας λένε χρειάστηκε να δράσουμε επιγόντως. Μα σήμερα είμαστε ακριβώς τριμωγμένοι στον τοίχο. Για ποιο λόγο. Ε, γιατί όλες αυτές οι επιλογές που κάναμε αυτόν τον καιρό ήταν ε, βράχυπρόθεσμες, κοντόφθαλμες. Η ίδια ευρωπαϊκή ιδέα κινδυνεύει, απειλείται. Εμείς είμαστε η πρώτη φωνή της Ευρώπης, γιατί εκπροσωπούμε τους λαούς της Ευρώπης. Έχει έρθει η ώρα να ακούσετε τη φωνή του Κοινοβουλίου. Ε, για ένα λεπτό, ο κύριος Τζαμπάσκι. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ε, ε, συμφωνούμε ούτε με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ούτε με το σχέδιο ανάκαμψη, γιατί αντιβαίνουν στις διατάξεις των ευρωπαϊκών συνθήκων. Εσείς ε, είστε υπέρμαχοι δήθεν του κράτους δικαίου, αλλά δέχεστε τέτοιε προτάσει που αντιβαίνουν στη συνθήκη. Δανείζεστε στι πλάτε των παιδιών μας, χωρί να ζητάτε τη γνώμη μα, ενώ ε, τα παιδιά μα θα πρέπει να αποπληρώσουν τα δάνειά σα. Και επίση ε, θα διανύμουμε τα κονδύλια αυτά του κοινού δανείου με τη μορφή δανείων και με τη μορφή επιχορηγήσεων. Ε, μα ε, έτσι εφαρμόζουμε τις αρχές του κομμουνισμού με αυτή την αμοιβεοποίηση και ξέρετε ποια, ποιο ήταν το τέλος του κομμουνισμού, που κατέληξε. Μιλάτε και τάχα κόπτεστε για το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου προβλέπει έναν εξάρτητο δικαστικό σύστημα. Μην προσπαθήσετε να αλλάξετε την κοινωνία, μην προσπαθείτε να αλλάξετε το οικογενειακό δίκαιο. Κύριε Φοντερ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, θα πρέπει να αντλήσετε τα συμπεράσματα και να δαχθείτε από το παρελθόν. Γιατί δημιουργείται μια σοσιαλιστική Ευρώπη χωρίς μέλλον. Ο κύριος Μπελαμή. Κυρία Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο δεν δέχεται αυτή τη συμφωνία. Αυτά ήταν τα λόγια του άρθρου 3 που ψηφίσαμε σήμερα. Βέβαια, η αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών χωρών ήταν αναμενόμενη απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή κρίση και το σχέδιο ανάκαμψης δίνει κακές απαντήσεις σε μια ουσιαστική κρίση. Έχουμε την ε, κοινή χρέωση, τον κοινό δανεισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί μιλούν για ιστορική στιγμή μετά την πανδημία που έφερε πένθο και μια ανήκουστη πρωτοφανή οικονομική κρίση ω επίπτωση αυτή τη πανδημία. Και γι' αυτό δεν χαιρόμαστε. Κανείς δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να μετατρέψει τη τραγωδία αυτή σε μια ανέλπιστη ευκαιρία για να αναβιώσει παλιές ψευδεστήσει τις οποίες έχουμε επανειλημμένως πει όχι. Τι θα πούν οι πολίτες όταν διαπιστώσουν ότι το σχέδιο ανάκαμψης είναι ένα φεντεραλιστικό άλμα που απλώς δεν λέει το όνομά του ε, όταν συνειδητοποιήσουν ότι αυτός ο περιττός δανεισμός γιατί οι χώρες μας έχουν πρόσβαση στις χρηματαγορές έχουν ένα τμήμα που δεν τους αποκαλύπτουν οι κυβερνήσεις γιατί οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να αποπληρώσουν ένα, ένα χρέος που ηρωνικά έχει συναυτεί στο όνομά τους και δεν θα ξέρουν πώς θα το επιστρέψουν. Και γι' αυτό θυσιάσαμε ουσιαστικά, γι' αυτό το άλμα, μια Ευρώπη που χρειαζόμαστε. Θέλουμε επισητιστική ασφάλεια και παρόλα αυτά 40 δισεκατομμύρια κόβουμε από την κοινή γεωρική πολιτική. Θέλουμε στρατηγική ανεξαρτησία και το Ταμείο Άμυνα χάνει το μισό προπολογισμό. Το θέμα της, ε, το Ταμείο Δική Μετάβαση από 30 πάει στα 10 δισεκατομμύρια. Και ενώ η υγειονομική κρίση έδειξε τι αδυναμίε μα, χάσαμε 13 δισεκατομμύρια και το, το πρόγραμμα για την υγεία από 9 στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ε, μόνο χρέη δημιουργούμε με τη συμφωνία αυτή. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε το μέλλον αναπροσανατολίζοντα σε ριζικά τι πολιτικέ μα και να προσαρμόσουμε την πολιτική ανταγωνισμού για να ξαναχτίσουμε τι οικονομίε μα και επιτέλου να αποφασίσουμε για το φόρο αναπροσαρμογή του άνθρακα που δεν έχουμε ε, καταλήξει στην αποτελεσματικότητά του. Αυτά θα πρέπει να πούμε τώρα, αντί να αναβάλουμε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον. Αυτά θα επιτρέψουν την πραγματική ανάκαμψη και θα πρέπει με αυτό να ασχοληθούμε ήδη από τώρα. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο ο κύριος Μπέλκα. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σήμερα συζητούμε το πώς ε, αντιδρά στις ε, σημερινές προκλήσεις, την πανδημία και τις μελλοντικές, ε, τη φορολογία, τους ιδίους πόρους, τον κοινό προϋπολογισμό. Και μιλάμε για κάτι ακόμη πιο σημαντικό, κέριο για την ύπαρξη της Ένωσης, για τις αξίες που θα έπρεπε να μας ενώνουν. Στην πατρίδα μου την Πολωνία το θέμα της ε, τήρησης του κράτους δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών συζητήσεων. Από τους κυβερνητικούς κύκλους ακούμε ότι ε, η, η τήρηση του κράτους δικαίου είναι, έχει διάμεσο ρόλο και ουσιαστικά έχει μείνει κενό γράμμα. Θέλουμε συγκεκριμένες αποφάσεις από το Συμβούλιο και όχι απλά λόγια. Γιατί στο Συμβούλιο ισχύει η αρχή για τα θέματα της διακυβέρνησης πλέον της ενισχυμένης πλειοψηφίας, αλλά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, λόγω των αρχών της ομοφωνίας, η Πολωνία θα βάλει βέτο σε αυτά τα θέματα. Και ταυτόχρονα η Πολωνία υπερασπίζει την κυριαρχία της, οπότε θα μπορούσε τιμόρυτα να παραβιάζει τις αρχές του κράτους δικαίου. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν. Είναι λοιπόν το αφήγημα αυτό σωστό και ακριβές. Γιατί μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και μερικές φορές φαίνεται ότι παρακάμπτουμε την αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να πούμε όχι μόνο στους Πολωνούς αλλά και σε όλους τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Μπέρ για ένα λεπτό. Κυρίες ε, Πρόεδροι, αγαπητέ Αλμισέλ, η Ευρώπη για να απογειωθεί χρειάζεται έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό που θα βοηθάει τη μεσαία τάξη, την καινοτομία, την εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς όμως αυτές οι πτυχές ε, περιεκόπησαν ε, και εδώ πέρα πρέπει ακριβώς να υπάρξει μια βελτίωση. Ειδικά δε τα κονδύλια για μια Ευρώπη τεχνολογικά προηγμένη με γεωπολιτική φύση έχουν πάρα πολύ μικρό προϋπολογισμό Γιατί παραμένουμε στα κεκτημένα, που είναι η φιλοδοξία, που είναι το θάρρος για να κάνουμε κάποια μεταρρύθμιση για το μέλλον. Πώς θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης για να έχουμε ευημερία. Όχι κύριε και κύριοι, πρέπει να το ξαναδούμε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα τα καταφέρουμε έτσι εις βάθος χρόνου. Αυτή λοιπόν είναι και η σωστή σχέση μεταξύ ε, επιδοτήσεων και δανείων. Λοιπόν, για αυτό το οποίο είπατε αγαπητέ συνάδελφοι, ναι, περισσότερες πληρωμές, αγαπητέ συνάδελφε, λιγότερες επιστροφές, λιγότερα δώρα. Περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Αυτό χρειάζεται η Ευρώπη για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή χρήση αυτών των κοινών χρεών που αναλαμβάνουμε. Για 1,5 λεπτό, ε, λεπτό κύριος Ρινάλντι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ιταλία τα τελευταία 20 χρόνια έχει συνεισφέρει συνολικά 160 δισεκατομμύρια καθαρά στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απλά κάνοντας μια πρόσθεση και στα διάφορα ταμεία. Όσο βεβαίως ε, κάνει όποιος βλέπει τα πράγματα αντικειμενικά και χωρίς ε, ιδεολογικές παροπίδες βλέπει ότι η Ιταλία στο τέλος του προγράμματος Next Generation όταν λάβουμε υπόψη και τις επιστροφές θα συνεχίσει να είναι καθαρός εισφορέας με αντίτιμο το να κατασφάξει φορολογικά τους πολίτες της οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται χωρίς καμία ελπίδα. Έχουμε λοιπόν παρά τα όσα λέγονται για την ε, Ιταλία καταλήξαμε να είμαστε καθαροί εισαγωγής. Λοιπόν, θα πρέπει πρώτα απ' όλα ε, όσοι μιλάνε να πλένουν καλά το στόμα τους, να έχουν κάνει καλά τους λογαριασμούς τους και μετά να μιλάνε για την Ιταλία. Ποιος θα πληρώσει λοιπόν όλα αυτά τα χρέη του προγράμματος Next Generation. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Going για ένα λεπτό. Ε, παρακολούθησα και εγώ την ε, Σύνοδο Κορυφής, όπως και εσείς, ε, το Σαββατοκύριακο. Έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα και μας λένε ότι δεν θα μπορέσουν τα ευρωπαϊκά κρατημέλη να έχουν το βάρος να αντιμετωπίσουν την κρίση στον 21ο αιώνα. Ο συμβασμός αυτός Εντάξει, έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Τα αρνητικά βεβαίως το είπαν αρκετοί. Είναι οι διάφορες περικοπές που έγιναν ειδικά στις πτυχές εκείνες του προπολογισμού που αφορούν το μέλλον. Η Ευρώπη θα πρέπει να απευθύνεται στους ανθρώπους και χρειάζονται πολύ περισσότερα σε αυτή την πτυχή Δεν ξέρω λοιπόν εάν μου διέφυγε εμένα το χειροκρότημα προς ανθρώπους οι οποίοι όντως δουλεύουν στον τομέα της υγείας, ε, στις οικογένειες, που ενισχύονται. Δεν βλέπω τίποτα σχετικό στον προϋπολογισμό. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει επιγόντως μια βελτίωση. Το οφείλουμε στους πολίτες της Ευρώπης. Αλλιώς πηγαίνουμε προς μια κατεύθυνση στην οποία δεν θέλουμε. Δηλαδή ο κόσμος νιώθει ότι δεν ε, τους κάνει κάτι καλό. Λοιπόν, πρέπει να ενισχυθούν άρα οι οικογένειες οι οποίες υπέφεραν στην κρίση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μισελ ζήτησε να παρέμβει τώρα γιατί ε, πρέπει να αναχωρήσει και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τις διάφορες τοποθετήσεις σας. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλο το Κοινοβούλιο ε, για το ρόλο που έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ως οραματιστή στο τελευταίο διάστημα. Θέλω να απαντήσω σύντομα σε κάποια σχόλια. Το πρώτο που θέλω να τονίσω και σημειώστε το είναι η αποφασιστικότητα που έχουμε αυτή τη φορά να δράσουμε γρήγορα και να δράσουμε δυνατά. Θυμόμαστε όλη τη χρηματοπιστωτική κρίση που έδειξε ότι όταν καθυστερούσαμε και δρούσαμε με τρόπο πολύ αδύναμο, ο λογαριασμός αυξανόταν. Λίγες εβδομάδες μόνο μετά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θελήσαμε να πείσουμε 27 ηγέτες που λογοδοτούν στα εθνικά τους κοινοβούλια να προχωρήσουμε. Και τολμώ να πω προς μία ε, αλλαγή ε, του ευρωπαϊκού μοντέλου τύπου Κοπέρνικου. Δηλαδή ε, με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, με το Ταμείο Ανάκαμψης αλλάζει τελείως ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση στοιχίζεται και προχωρεί. Είπατε ότι είναι παλιά αυτή η πολιτική συζήτηση, δεν είναι νέα, αλλά τούτη εδώ τη φορά κάναμε ένα απολύτως ουσιαστικό βήμα πρόοδου και χαίρομαι που θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εκεί γιατί υπάρχει ε, το θέμα των ε, τελών ή των φόρων για τον άνθρακα, ε, για τα ψηφιακά, για διάφορα άλλα θέματα. 450 εκατομμύρια πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη δημοκρατική διαδικασία και το δημοκρατικό γίγνεσθε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω επίσης να σας πω ότι αυτή η ενέργειά μας τώρα δεν είναι κατάληξη. Είναι αφετηρία ε, χρειάζεται πολλή δουλειά, πολλή ενέργεια, πολλή κινητοποίηση για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε αυτή τη συμφωνία που είναι στα χαρτιά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα γίνουν συζητήσεις ε, με πάθος και πολύ ενδιαφέρουσες στα Εθνικά Κοινοβούλια να μεταφραστεί λίγο στην πραγματική ζωή. Το είπα και εισαγωγικά και το επαναλαμβάνω. Δεν είναι απλώς θέμα χρημάτων, είναι θέμα αξιών, θέμα αρχών και προσανατολισμών που θέλουμε να δώσουμε στο ευρωπαϊκό εγχείρημα που μας κινητοποιεί και είναι μοναδικό, χωρίς προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία, 27 διαφορετικές χώρες, 450 εκατομμύρια που συνδέονται γύρω από κοινέ αξίες και φιλοδοξίες να προχωρήσουν έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο ανθρωπισμό ε, που να μοιραζόμαστε. Και τελευταίο, ακούω, ακούω υπερβολές. Ε, άκουσα και κάποια λόγια έτσι ε, λίγο αξιοθρύνητα εξερμιστικών κομμάτων που εκπροσωπούνται εδώ. Το κατανοώ. Επιλέγετε την αναδίπλωση, επιλέγετε το μίσος, επιλέγετε το διαχωρισμό, επιλέγετε την απόρριψη. Εμείς επιλέγουμε την ανοχή, το άνοιγμα και για σας είναι θλιβερή ημέρα, ενώ για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους είναι μια μέρα χαράς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την συμμετοχή σας ε, σήμερα στην ε, έκτακτη αυτή συνεδρίαση. Επιστρέφουμε στις ε, παρεμβάσεις των βουλευτών. Κύριε Ράγκελ, έχετε τον λόγο για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και επιτρέψτε μου να πω συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Μισελ και στο Συμβούλιο για αυτή την ιστορική συμφωνία. Αλλά είναι ηρωνικό ότι τώρα που επιτέλους έχουμε πραγματικά ευρωπαϊκά κονδύλια θα τα δαπανίσουμε κυρίως σε εθνικούς φακέλους, σε εθνικούς προϋπολογισμούς, εθνικά προβλήματα και όχι σε πανευρωπαϊκά μεγαλεπίβολα προγράμματα. Η σοβαρότατη κρίση που περάσαμε στα υγειονομικά μας συστήματα, μια κρίση υγειονομική, θα πρέπει πρώτα να μας φέρει να αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα και στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Ταυτόχρονα όμως έχουμε μια σοβαρότατη οικονομική και κοινωνική κρίση και γι' αυτό είναι σημαντικό να πούμε ότι η συμφωνία όντως είναι ιστορική. Θέτει όμως ένα, ένα ερώτημα. Πώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν έχουν πια δικαιολογίες και προσχήματα. Έχουν τα μέσα να αντιμετωπίσουν την κρίση την κρίση που χτύπησε τους πολίτες, τι επιχειρήσεις, τους εργαζόμενου. Σε ό,τι αφορά τώρα το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, οφείλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου. Κρίμα που δεν έχουμε ένα μεγάλο επίβολο πρόγραμμα για την υγεία και κρίμα που ε, μειώνουμε το Erasmus Plus και την έρευνα. Και εμείς ε, θα ε, δεχτούμε το τα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο αν διορθούν αυτά τα προβλήματα. Μία σοσιαλίστρια Πορτογαλία μίλησε για τη διάσκεψη για το, μέλλον της Ευρώπης. Η Πορτογαλική κυβέρνηση δυστυχώς όμως ήταν αυτή που μπλόκαρε περισσότερο στο Συμβούλιο τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και μίλησε για τις αξίες και τα δικαιώματα. Αλλά ο Πρωθυπουργό Κώστα ήταν αυτός που ζήτησε απόλυτο διαχωρισμό μεταξύ του σχεδίου και του Ταμείου Ανάκαμψης και του κράτους δικαίου. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φριτζόν, για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σοβαρότατες προκλήσεις και θα πρέπει από κοινού να λύσουμε τις κρίσεις. Θέλουμε ένα σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που θα δίνει προτεραιότητα στην απασχόληση και στο κλίμα και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και ένα πακέτο ανάκαμψης για να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα κρίση. Και φυσικά έχουμε ανάγκη και από την ε, πράσινη μετάβαση. Και χαίρομαι που μετά από ε, τέσσερα μερόνυχτα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Συμβούλιο ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για το σχέδιο ανάκαμψης και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ιστορική πρόοδος άνευ προηγουμένου. Οι διαπραγματεύσεις προϋποθέτουν δούνε και λαβίν και φυσικά ε, η κατάσταση είναι διαφορετική στα κράτη-μέλη, όπως διαφορετική είναι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των Ευρωβουλευτών. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να υπομιστούν τις ευθύνες τους, και τα κράτη-μέλη και εμείς. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα πρωτοστατεί στην προσπάθεια μετριασμού των κλιματικών αλλαγών και θα προστατεύει την απασχόλησή της. Επίσης, θα πρέπει ταυτόχρονα να λαμβάνουμε υπόψη το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη, όχι σε 26, σε 25. Στις 27 χώρες μέλη θα πρέπει να σταθούμε υπέρμαχοι του κράτους δικαίου. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη για τις επερχόμενες γενιές. Γιατί το κάνουμε, εγώ το κάνω για τα παιδιά μου, για τα παιδιά των παιδιών μου και των μέλων τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πισλάρου για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κύριε Πρόεδρε, Φαντερ Λάιεν, αγαπητοί συναδελφοί, όλοι ακούσαμε το τι θέλουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα πρέπει να συζητήσουμε εμείς το τι θέλουν οι πολίτες. Συγκεκριμένα, ας ακούσουμε το τι θέλει η επόμενη γενιά. Γιατί το λέμε, αλλά δεν ακούμε. Βλέπουμε ε, προγράμματα όπως το Erasmus Plus, η ε, εγγύηση για την νεολαία, ψηφιακή Ευρώπη, περικόπτονται. 90% των κονδυλίων για την επόμενη γενιά θα πάνε στο Ταμείο Ανάκαμψης, το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να νεωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως συνεισηγητής επί του θέματος θέλω να δεσμευτώ για κάτι. Το μέσο ανάκαμψης θα είναι μέσο για την επόμενη γενιά θα ζητήσω να υπάρξει ένας πυλώνας σχεδιασμένος ειδικά για την νεολαία και για τα παιδιά. Θα προετοιμάσουμε το μέλλον μόνο εάν βοηθήσουμε την επόμενη γενιά. Όχι μόνο να τους φορτώσουμε το λογαριασμό, αλλά να έχουν και φωνή για τα παιδιά μας, για την νεολαία μας. Το κοινοβούλιο θα είναι η φωνή σας. Σας ευχαριστώ. Ζλοτόφσκι, παρακαλώ για ένα λεπτό. Με μικρόφωνο όμως. Ε, κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε δύσκολο συμβιβασμό για το νέο προϋπολογισμό ένα προϋπολογισμός που είναι απαραίτητο για την ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή Οικονομία μετά την κρίση που μα έπληξε. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντε ε, να επενεθούν, όλοι αξίζουν συγχαρητηρίων, όπω είπε και ο Πρωθυπουργό ε, Μοραβιέτσκι. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία. Βέβαια, ακούστηκαν και επικρίσεις μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι υπερβολικές όμως και δείχνουν και μια υποκρισία. Θα ήθελα να πω ε, στους συναδέλφους και τους Πολωνούς που ε, αναφέρουν τον μηχανισμό κράτους δικαίου, την απόπειρα δημιουργίας ε, μηχανισμού εκτός συνθήκων για τον έλεγχο του κράτους δικαίου. Δεν στηρίζει το μηχανισμό αυτό σε πραγματικά περιστατικά, αλλά στη συμπάθεια την αντιπάθεια που προκαλούν μερικές κυβερνήσεις. Όλα τα όλα συνέες διατάξεις της Πολωνίας ε, συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Πολωνία είναι κράτος δικαίου. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία. Μερικοί όμως στην αίθουσα θέλουν να εκμεταλλευτούν το μηχανισμό κράτος δικαίου για να ασκήσουν πιέσεις σε ε, πρωθυπουργούς ή κυβερνήσεις που δεν είναι της αρεσκίας τους. Η Πολωνία τηρεί τις συνθήκες ε, ε, και οι συνθήκες ε, θα πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο για το μηχανισμό του κράτους δικαίου. Και το Συμβούλιο σωστά τέτοια μήνυματα έδωσε. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην καταστρέψει το αποτέλεσμα των δύσκολων αυτών διαπραγματεύσεων που δημιούργησαν σημαντικέ προσδοκίε. Γιατί περισσότερο από ποτέ οι Ευρωπαίοι χρειάζονται σήμερα συνεργασία και όχι στήρε διαμάχε. Ευχαριστώ. ένα 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τις τελευταίες μέρες έγινε ένα τεράστιο βήμα προόδου. Πολιτική δεύσμευση των ηγετών για το Ταμείο Ανάκαμψης και προπολογισμό δισεκατομμυρίων. Μπορούμε έτσι να επενδύσουμε και πάλι στο ευρωπαϊκό μας μέλλον και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα τέτοιο Ταμείο Ανάκαμψης είναι πρωτόγνωρο από πλευράς τάξης μεγέθους. Το λεγόμενο Next Generation έχει 390 εκατομμύρια επιχορηγήσεις και 360 δισεκατομμύρια συγγνώμη, δάνεια. Και πάλι μπορούν να πάρουν μπρος λοιπόν τα κράτη-μέλη. Από την άλλη, ε, με βάση ε, τα δάνεια μπορεί κάθε χώρα να αποπληρώνει με βάση τη δυνατότητά της. Και ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Βέλγιο ε, είναι ε, χρήσιμο και αυτό που αποφασίστηκε για τον Brexit. Ε, θα πρέπει γρήγορα να επενδύσουμε στην έρευνα και την καινοτομία, να βρούμε γρήγορα εμβόλιο για τον κορονοϊό, να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο. Αυτά είναι προτεραιότητες. Επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη και στο πρόγραμμα των ορίζων είναι απολύτως απαραίτητα. Επίσης, οι μεγάλες περικοπές ε, στην υγεία και στην άμυνα με βρίσκουν απολύτως και κατηγορηματικά αντίθετο. Δεν μπορεί να έχει στρατηγική αυτονομία η Ένωση αν δεν συνεργαστεί. Τώρα περιμένουμε ε, όλο και περισσότερο ε, πιθανό είναι το σκληρό Brexit και ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού η συμφωνία για τον προπολογισμό μπορεί να βελτιωθεί και πρέπει να βελτιωθεί παρόλα αυτά και παρόλε τι διαπραγματεύσει. Η κυρία Γιονγκέριου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χώρα μου στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες δεν είχε την καλύτερη ε, εικόνα. Ηγέτης των τεσσάρων φιδωλών. Αυτό έχει να κάνει ε, με ε, τον Πρωθυπουργό Ρούτε. Αν κυβερνούσε το δικό μας εργατικό κόμμα θα ήταν τελείως διαφορετικά ε, τα πράγματα. Ε, είναι καλό για τους Ευρωπαίους, είναι καλό για την ενότητα, είναι μεγαλύτερη ισχύ της Ευρώπης και απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Παρ' όλα αυτά, ο προϋπολογισμός αυτός είναι το ίδιο παλιό κρασί σε νέα μπουκάλια. Ε, οι νέες προτεραιότητες ε, ε, για τους νέους, για την ανεργία των νέων, για την υγεία, για το περιβάλλον. Φαίνεται μια χαμένη κρίση, ακριβώς στα μέση του κορονοϊού και δεν έχω πει τίποτα ακόμα για την ασθενή σύνδεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με το κράτος δικαίου. Πραγματικά, Πρόεδρε, είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά μόλις τώρα ξεκινήσαμε. Eh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μας δημιουργεί την ελπίδα ότι θα βγούμε ενισχυμένοι από αυτή την κρίση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες διεκπαιρέωσαν το ρόλο τους και αξίζουν επένων και ευγνωμοσύνης. Όλα τώρα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και να στηρίξουν αυτή τη συμφωνία που είναι σημαντική για το ευρωπαϊκό κοινό. Ω συντονιστή από την Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη, δεν θέλω να μειωθούν τα κονδύλια του Ταμείου Δίκαιη Μετάβαση. Το αντίθετο, μάλιστα. Θα ήθελα να ενισχυθεί η πολιτική συνοχή και χαιρετίζω τη σχετική πρόταση, γιατί η πολιτική συνοχή δημιουργεί νέε θέσει εργασία. Ευχαριστώ την Επίτροπο Φερέιρα, που είναι αρμόδια για τη συνοχή. Την ευχαριστώ για το έργο της, αξιέπαινο ε, και θα ήθελα να πω εγκατακλείδη ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, που θα χρησιμοποιηθούν για τα κλιματικά μέτρα θα πρέπει να είναι ε, ανοιχτά σε όλες τις νέες τεχνολογίες και στην πυρηνική. Σας ευχαριστώ. Ρέσλερ για ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Με μικρόφωνο όμως. Ναι, τώρα δουλεύει. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τη στιγμή μιας ε, πρωτοφανούς υγειονομικής και οικονομικής κρίσης και μετά από μια δραματική, τραγική άνοιξη, ασυνήθιστο καλοκαίρι και αβέβαιο φθινόπωρο, επιτέλους ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε ένα θετικό μήνυμα το μήνυμα της ευθύνης και της συνεργασίας στην Ευρώπη. Ένα μήνυμα που χρειαζόμαστε σήμερα στην Ευρώπη. Κάποιες χώρες, ε, οικονομικοί κλάδοι αλλά και γενιές επλήγησαν περισσότερο από άλλους και γι' αυτό ε, είναι θεμελιώδους σημασίας ε, να αποτρέψουμε την εμβάθυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Για την πατρίδα μου την Κροατία, αλλά και για ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η απτή αλληλεγγύη δίνει μεγάλη ευκαιρία για την οικονομική ανάκαμψη και την ενίσχυση με την ψηφιακή ταυτόχρονα μεταρρύθμιση και τον ε, ε, περιβαλλοντικό μετασχηματισμό. Αυτό είναι απόλυτη προπόθεση και για τι μελλοντικέ γενιέ. Και επίση είναι σαφέ ότι βρισκόμαστε στην αφετηρία αυτή τη συζήτηση. Και το σχέδιο ανάκαμψη και το Ταμείο Ανάκαμψη ε, ε, με τι μαζικέ αυτέ επενδύσει ε, μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά προγράμματα. Αλλά και η έρευνα και η ψηφιακή Ευρώπη και η παιδεία είναι σημαντική κλάδη για το μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο με ερετά αιρετούς εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών ε, μπορεί με τις συζητήσεις να συμπληρώσει αυτή την καλή συμφωνία και να της δώσει μια ισχυρή ευρωπαϊκή προοπτική, βελτιώνοντας τη συμφωνία αυτή. Θα πρέπει επίσης να δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει κάποια ιστορικά βήματα όταν κάτι τέτοιο ε, είναι απαραίτητο για όλες τις γενιές και για όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βόντερ Λάιν, περισσότερα χρήματα για την υγεία, το κλίμα και την απασχόληση χωρί ε, επιβάρηση των κρατικών προϋπολογισμών. Καλό ο ψηφιακό φόρος, αλλά είναι δύο δι ετησίω. Ε, ε, Φόρο στα πλαστικά φανταστικά, αλλά είναι πέντε δι και θα μειωθούν. αυτή η καλύτερη λύση που θα μπορούσε να φέρει περισσότερα χρήματα και να συμφωνήσουν περισσότερες χώρες ήταν το τέλος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το συζήτησε το Συμβούλιο και μπράβο το λέει στα συμπεράσματα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται συμφωνία και μάλιστα τώρα παρά την κρίση θα μπορούσε να φέρει 50 δις. Το 2011 η Επιτροπή Μπαρόζο είχε προτείνει σχετική οδηγία και παρά το Brexit και την κρίση μπορεί να φέρει αυτό 50 δις ετησίως. Αυτό είναι 15 δις για το χρέος και 35 δις για την υγεία, το κλίμα και την απασχόληση. Αυτό ζητούν οι σοσιαλδημοκράτες. Εδώ η λύση για ένα πιο φιλόδοξο προπολογισμό χωρίς δεκάρα από τα κράτη-μέλη. Είπε το Συμβούλιο ότι είναι προτεραιότητα και η Γερμανία και χαίρομαι Είμαι, είμαι για το προπολογισμό του 2021. Αλλά ως πολίτης και ως βουλευτής δεν θα δεχτώ προπολογισμό αν δεν υπάρξει συμφωνία για το φόρο χρηματοστατικών συναλλαγών. Θέλουμε αυτά τα 500 δις επιπλέον. Σας ευχαριστώ. Ινετφέλντ παρακαλώ. Σοφία για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω την παρέμβασή μου θα ήθελα να πω ότι είναι λυπηρό το ότι η ηγεσία της ε, Κομισιόν και του Συμβουλίου συνηθίζουν να φεύγουν πριν από το τέλος της συζήτησης. Για μια τόσο σημαντική συζήτηση ε, θα περίμενα να παραμείνουν μέχρι το τέλος. Συνάδελφοι, σήμερα έχουμε γενέθλια είναι τα γενέθλια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και στην Συνθήκη των Παρισίων του 1959 δόθηκε στην Υπατιαρχή η δυνατότητα να επιβάλλει φόρους ε, και να δανείζεται λεφτά. η δε αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονταν με πλειοψηφία. Τότε είχαν το όραμα η σημερινή συζήτηση δεν αφορά τα λεφτά και τους αριθμούς. Αφορά το πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε την ευρωπαϊκή μας κοινωνία. Αφορά την επιλογή μεταξύ της παλαιάς και της νέας Ευρώπης. Επιστροφές είναι η παλιά Ευρώπη του 1984. Επένδυση στην έρευνα στο κράτος δικαίου και την κλιματική αλλαγή είναι η νέα Ευρώπη. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι Ευρωπαίοι άνω των 200 εκατομμυρίων μα έδωσαν μια εντολή σε ευρωεκλογέ. Είχαν προσδοκίε για το μέλλον. Το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία και έχουμε καθήκον να την χρησιμοποιήσουμε. Α κάνουμε λοιπόν αυτό το βήμα προ τα εμπρό. Σα ευχαριστώ. Έχετε δίκιο βεβαίω ε, με την παρατήρησή σα, ε, ε, η οποία θα διαβιβαστεί. Νόβακοφ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, εκπρόσωποι του Συμβουλίου, είπαν ε, πολλοί συνάδελφοι που έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρατε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτό το οποίο καταφέρατε τουλάχιστον μετά από πέντε μέρες. Σίγουρα η συμφωνία δεν είναι τέλεια και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να την κάνει τέλεια. Ορισμένες από τις ε, υποσχέσεις μας προβληματίζουν. Πώς θα βγούμε από την κρίση και ταυτόχρονα θα μειώσουμε ε, τις ε, δαπάνες για την υγεία πώς ε, θα βελτιώσουμε το κλίμα ενώ περικόπτονται τα ταμεία για τη δίκαιη μετάβαση. Εμείς αγωνιστήκαμε για να αυξηθούν οι πόροι ε, του προγράμματος Έρασμος. Τελικά έχω την αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ε, έχει μεγαλύτερο νόημα. Περιμέναμε πάνω από 600 ημέρες για να έρθει αυτή η συμφωνία και τώρα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη βελτιώσουμε. Κάθε βράδυ που λέμε καληνύχτα στα παιδιά μας, τους υποσχόμαστε ένα καλύτερο αύριο και ότι όταν θα ξημερώσει θα τους πούμε και καλημέρα. Ε, αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε. Κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν επιτρέπεται να μειώσουμε την πολιτική συνοχή. Αυτά περιμένουν από εμά οι πολίτες, από το Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο υπάρχει για τους πολίτες του. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη με το Ταμείο Ανάκαμψης ξανααναλαμβάνει τα ενία του μέλλοντό τη. Ε, Κοινή φόρη, κοινό χρέο, για να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέλλον. Έτσι φτιάχνουν το μέλλον του οι αυτή τη φορά οι μεταρρυθμίσεις ε, θα είναι υπέρ των Ευρωπαίων, θα επενδύουν στους Ευρωπαίους, θα επενδύουν σε μια πιο ανταγωνιστική, πράσινη, ψηφιακή οικονομία με ποιοτικέ θέσει απασχόλησης. Είμαστε υπέρ μια πιο ανθεκτική βιομηχανία Και φυσικά ε, μια ανάπτυξη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς που θα εντείνει τη σύγκληση. Μερικές φορές ε, διδα, έχουμε διδαχθεί από τα παθήματα του παρελθόντος. Δεν θα διασώσουμε κάποιες χώρες, αλλά την ίδια την Ευρώπη. Και με φιλοδοξία και αλληλεγγύη θα το καταφέρουμε. Μας κόστησε πολύ αυτή η συμφωνία. Συμβάλαμε και εμείς και πολλές κυβερνήσεις όπως η Ισπανική. Αλλά το τίμημα ήταν πολύ υψηλό. Μία ατυχής λυπηρή πρόταση ε, για, την τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και γι' αυτό απαιτούμε, ως συναρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, απαιτούμε έναν κοινοτικό προϋπολογισμό που θα είναι στο ύψος των ε, προκλήσεων και θέλουμε ε, χρηματοδότηση που θα συνάδει με τα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Η κυρία Ελίδια Περέιρα τώρα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, πριν από 7 μήνες ξυπνήσαμε σε μια νέα πραγματικότητα. Είδαμε η διεισόμαση την καταστροφική επέλαση ενός άγνωστου μέχρι πρώτη νοσίου και την εξάπλωση του παγκοσμίω με ταχύτητα εφάμιλη του φόβου που προκάλεσε. Η μία μετά την άλλη. Όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επλήγησαν από τον ιό αυτό, από τον κορονοϊό και όλες χωρίς καμία εξαίρεση θρύνησαν πολλά θύματα ο φόβος και η ανάγκη να αναχαιτήσουμε τον ιό ε, έκλεισαν τα εργοστάσια μας, τα σχολεία μας ε, και άφησαν μετέωρη τη ζωή μας για πολλούς μήνες. Αλλά η Ευρώπη δεν σταμάτησε και για μια ακόμη φορά στάθηκε στο ύψος των προκλήσεων και έκλεισε το στόμα με δράση και αποφάσεις στους λαϊκιστές που συνεχώς αναγγέλουν το τέλος, τη συντέλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι με την πρόταση για τον φόρο για τα πλαστικά ω νέο ίδιο πόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα μικρό βήμα, αλλά με μεγάλη σημασία για τις νέε γενιέ. Βέβαια δεν είναι όλες οι ειδήσει ε, χαρμόσυνες. Το Συμβούλιο δυστυχώς ε, ε, απαρνήθηκε το μέσο για την αφαιριότητα των επιχειρήσεων ε, που είναι σημαντικό, σημαντική βοήθεια έκτακτη ανάγκη και συμφώνησε σε περικοπές στο ορίζοντα 2020 στο πρόγραμμα Έρασμο και στο Ταμείο Δικής Μετάβασης. Και δυστυχώς ε, ε, ο ωραίος τίτλος Next Generation EU, η Ευρώπη τη νέας γενιάς χάνει την σημασία του. Ο φιλόσοφος, ο Βάσκος φιλόσοφος Δανιέλ Ναρίτη είπε ότι πολλές φορές το μέλλον είναι ο κάλαθος αρχή, χρήστων του παρόντος. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, ανησυχούμε ιδιαίτερος για τι διεθνεί μα ευθύνε. Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει τίποτα για ανθρωπιστική βοήθεια και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο έχει περικοπεί στον τομέα της αναπτυξιακή συνεργασίας. Η αλληλεγγύη υποφέρει ειδικά σε μια στιγμή στην οποία οι εταίροι μας την έχουν μεγάλη ανάγκη. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Οι σοσιαλδημοκράτες εργάζονται για μια επέκταση του υφιστάμενου προγράμματος για καλές δουλειές και για οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε ήδη θέση της ε, Σχετικέ ε, προτεραιότητε σε Γερμανία και Ευρώπη. Αλλά ένα είναι σαφέ. Οι πολίτες σε Βαρσοβία και ε, Βουδαπέστη δεν έχουν κάποια τιμή. Δεν εξαγοράζονται ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε την μέρα στην οποία θα γίνει η ψηφοφορία για το ΠΔΠ. Σας ευχαριστώ κύριε Κάρας. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Κυρίες και κύριοι, ο συμβιβασμός του Συμβουλίου είναι η αρχή των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι αναγκαίες γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε την επανεθνικοποίηση, το ότι δεν υπάρχει κάποια ε, κάποιος προγραμματισμός ε, για το μέλλον έτσι απλά. Θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ε, ATM, ούτε είναι παζάρι. Είμαστε μια κοινότητα δικαίου. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Θέλουμε να είμαστε μια κοινότητα που κοιτάει προς το μέλλον και είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο μέλλον, όχι ε, απέναντι στα κόμματα και τον λαϊκισμό, τον δεξιό και τον ε, εθνικιστικό. Και αυτά τα οποία μας λέει εδώ πέρα ο κύριος Μισελ είναι διαφορετικά από την επικοινωνία της ιστορικής συμφωνίας των 750 δισεκατομμυρίων και τα όσα λένε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στις χώρες γιατί δεν συμπεριφέρονται με ευρωπαϊκή ευθύνη αλλά συμπεριφέρονται με εθνικό λαϊκισμό. Πρέπει να πω επίσης κάτι ξεκαθαρό εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα δεχτούμε αποφάσεις χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξουν λεφτά για όσους παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές αξίες μας. Ούτε περικοπές στην έρευνα, κλίμα, επενδύσεις και κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει να υπάρξει εισαγωγή ενός μηχανισμού κράτους δικαίου και ένα σχέδιο αποπληρωμής με ουσία θα πρέπει να μην υπάρχει ομοφωνία για να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Άγγελ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η επίτευξη συμφωνίας και απάντηση σε μια πρωτοφανή κρίση στην Ευρώπη είναι θετικά χαρμόσυνα, είναι η ιστορική συμφωνία, αλλά μόνο το τμήμα που αφορά το μείον άκαμψη, το Next Generation EU, που έχει ένα μεγάλο τμήμα επιχορήγηση και κοινό δανεισμό, κοινό ευρωπαϊκό χρέο. Αυτό είναι αλληλεγγύη και καλύτερη απάντηση στην κρίση από το 2008. Σε ό,τι αφορά όμω το PDLTP, που υποτίθεται θα κάνει την Ευρώπη πιο ανθεκτική, πιο κοινωνική, πιο σύγχρονη, πιο φιλοπεριβαλλοντική, για τις επόμενες γενιές ε, δεν είναι και πολύ καλές ειδήσει για τις επόμενες γενιές, ούτε είναι ιστορική συμφωνία για το ΠΔΠ. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεχτεί περικοπές σε προγράμματα που στρέφονται προς το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ε, συμφωνούμε με την άβληση του κράτους δικαίου και γι' αυτό στο ψήφισμα θέλουμε να προσθέσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία. Και κρίμα που δεν καταργήθηκαν και τα rebates, οι επιστροφές. Εδώ το Συμβούλιο έχασε μια ευκαιρία να μας βγάλει από τη συζήτηση για τον καθαρό συνεισφορέα. Η Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από απλές και σήμερα εμείς ως Ευρωβουλευτές που είμαστε οι μόνοι άμεσα εκλεγμένοι στο άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο, θέλουμε να εγκρίνουμε το ψήφισμα καλωσορίζοντας και χαιρετίζοντα το Ταμείο Ανάκαμψη, αλλά λέγοντα ότι το ΠΔΕΛΤΑΠΗ δεν είναι αρκετό. Δεν επαρκεί ούτε από οικονομική άποψη, αλλά ούτε και προ την προστασία του δικαίου και της και της αξίας. Δεν ε, θέλουμε να καταπιούμε πικρά χάπια. Αξίζουμε περισσότερο. Κύριε Σπυράκη. τη Ευρωπαϊκή Ένωση έκαναν ένα ιστορικό βήμα εγκρίνοντα κοινό δανεισμό για να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη ύφεση από τον πόλεμο. Είναι τώρα ανάγκη οι πόροι αυτοί να συντονιστούν προκειμένου η ενιαία αγορά και οι οικονομίε μα να είναι περισσότερο πράσινε, περισσότερο ψηφιακές και περισσότερο ανθεκτικές βεβαίω αυτό το ιστορικό βήμα βασίζεται σε έναν ιστορικό συμβιβασμό από τον οποίο εμεί ως κοινοβούλιο δεν μπορούμε να δεχτούμε την αποσύνδεση της χρηματοδότηση από το κράτο δικαίου τη μείωση των κονδυλίων για την έρευνα την υγεία και την παιδεία τη μείωση των κονδυλίων για το ταμείο δίκαιης μετάβασης που τόσο χρειάζονται οι περιοχές της δυτικής μακεδονίας και της μεγαλόπολης. ελπίζουμε ότι αυτά θα αλλάξουν στη διαπραγμάτευση. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αυτές τις ώρες στη μεσόγειο εξελίσσονται σκηνές πρωτοφανούς έντασης με ευθύνη τη τουρκίας. η τουρκία μια υποψήφια χώρα για ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελλάδος έχει εκδώσει ναύτεξ με στόχο να κάνει σεισμικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα της ελλάδος η τουρκία παραβιάζει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της κύπρου η τουρκία προκαλεί τη γαλλία η τουρκία παραβιάζει το εμπόριο των όπλων στη λιβύη προσβάλλει τις αξίες του δυτικού πολιτισμού μετατρέποντας το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς την αγία σοφία σε τζαμί. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ζητάμε τώρα να καταρτιστεί άμεσα ο κατάλογος των κυρώσεων της ευρωπαϊκής ένωσης κατά της τουρκίας. είναι ο μόνος τρόπος να στείλει η ένωση ένα σαφές και καθαρό μήνυμα ότι δεν ανέχεται να παραβιάζονται τα κυριαρχικά βασικά δικαιώματα των μελών τη ότι δεν ανέχεται απειλέ στα σύνορά τη εργαλειοποιώντα ανθρώπου που υποφέρουν. είναι η ώρα η ευρωπαϊκή ένωση να πάρει τη θέση που τη αναλογεί ω παίκτη στη διεθνή σκακέρα τη εξωτερική πολιτική. πλέον οποιαδήποτε ανοχή στην τουρκία υπονομεύει την ισχύ τη ευρωπαϊκή ένωση υπονομεύει το κοινό μα μέλλον. σα ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρέμβαση, κυρία το Συμβούλιο αυτό θα μείνει οπωσδήποτε στην ευρωπαϊκή ιστορία γιατί πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση για το μέλλον μας. Επιλέγουμε την ε, Ευρωπαϊκή Ενότητα, την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών για να δημιουργήσουμε κοινά μέσα. Λοιπόν, αυτά δεν είναι μόνο ζητήματα οικονομίας, ε, αφορούν την υγεία και την κοινωνική ψυχή της Ευρώπης. Και βεβαίως ε, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί κάθε χώρα πλέον να καταπέσει και αυτό σημαίνει ότι θα, αν πέσει μία θα πέσουν όλες. Ε, λοιπόν, Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν ε, και διάφορες ε, ψευδεστήσεις για τι έχουμε ένα πι δελτα πι το οποίο δεν έχει συνοχή και έχει αντιφάσεις. Δεν ε, το αντιλαμβάνουμε εγώ. Πώς μπορούμε να έχουμε περικοπές σε πολιτισμό κτλ. Δεν μπορούμε να μειώνουμε την, τον προπολογισμό για την έρευνα. Δηλαδή περάσαμε μήνες ε, και κρεμόμασταν από τα χείλη των επιστημόνων για να δούμε πώς θα επιζήσουμε και τώρα σήμερα ε, το ξεχνάμε. Μα η οικονομία, το μέλλον μα εξαρτάται από τις εμιλιολογίε που κάνουμε, από τα φάρμακα, από το οτιδήποτε. Έχουμε λοιπόν όλους αυτούς τους έρευνητέ ε, ε, που έχουν ανεπαρκείς επιδοτήσεις. Ε, θα σηκωθούν να φύγουν αν δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και εσάς δεν σας έχουν ευχαριστήσει αρκετά εντό αίθουσα ε, για τα αποτελέσματα. Σα ευχαριστώ τώρα για να απαντήσει εξ ονόματο ε, τη Κομισιόν ο Επίτροπο κ. Χάν. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, Υπουργέ, κυρίε και κύριοι. Καταρχά, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω ειλικρινά καρδιάς για την έκτακτη αυτή σύνοδό σας. Και κάποιοι από εσά ε, διακόψατε και τις διακοπές σας που τόσο ε, είχατε ανάγκη και κερδίσει. Έπρεπε όμως γρήγορα να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες. Έτσι κι αλλιώς διήρκησε αρκετά διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο ε, μέχρι να καταλήξουν σε κοινή θέση. Τώρα υπάρχει η κοινή θέση. Η κριτική σας για την περικοδότηση, ιδιαίτερα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, είναι βάσιμη ορισμένα μπορούν να ε, διορθωθούν στις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα εκείνοι οι τομείς που δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από το Next Generation. Σκέφτομαι εδώ, ας πούμε, την εξωτερική πολιτική. Εκεί ε, έχουμε εξηγήσει και επανειλημμένα συζητήσει και μαζικά πόσο σημαντικό είναι στην πολιτική γειτονία, στην Αφρική να είμαστε παρόντες, να δραστηριοποιούμαστε και στο παρελθόν και σήμερα εξακολουθούν να ισχύουν αυτά και για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Αλλά επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και σε άλλα ε, μέρη της γης να υπάρξουν, ε, εφόσον βρεθούν, και τα φάρμακα και τα εμβόλια για την πανδημία. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. Γι' αυτό ε, πραγματικά πιστεύω ότι σε αυτούς τους τομείς υπάρχει δυνατότητα ε, και περιθώριο βελτίωσης. Πολύ συχνά αναφερθήκατε στο κράτος δικαίου. Ε, η κυρία Πύρη νομίζω ήταν μία από εκείνους που είπαν ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Ε, προφανώς ο καθένας εμπιστεύει στην πατρίδα του και βλέπει αυτά που θέλει να δει. Αυτά όμως που μετράνε είναι αυτά που γράφονται στα συμπεράσματα και τελικά εγκρίνονται. Επομένως υπάρχει μια πολιτική δήλωση, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα να μεταφραστούν όλα αυτά σε νομοθετικές ρυθμίσεις και να και φυσικά θα είστε και εσείς τμήμα της συζήτηση αυτής και τελικά της απόφασης αυτής. Σε ό,τι αφορά τους ιδίους πόρους, θέλω να πραγματικά, πραγματικά να ευχαριστήσω για την ισχυρή σας υποστήριξη. Είναι προδιαγεγραμμένο αυτό το σχέδιο και ο δρόμος έπρεπε να δούμε ποια είναι η τάξη μεγέθους πρώτα απ' όλα για την οποία συζητούμε η οποία δεν θα πρέπει απλώς να συγκεντρωθεί από τις χρηματαγορές αλλά και να αποπληρωθεί. Ε, και ως ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα έχουμε να λάβει την εντολή να σχεδιάσουμε τις λεπτομέρειες. Τι είδους νέοι πόροι μπορεί να προκύψουν, μπορώ να σας δώσω κάποιες ενδείξεις Για το Κοινοβούλιο συμφωνούν είναι από τα συμπεράσματα ε, και θα πρέπει να κάνουμε μια καλή αξιολόγηση. Ε, ορισμένες πηγές εσόδων μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν ταχύτερα. Κάποια άλλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο γιατί έχουν μεγαλύτερη περιπλοκότητα. Ε, ας πούμε ο φόρος ή το τέλος ή ο μηχανισμός επιστροφής στα σύνορα για το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό είναι ένα θέμα δύσκολο και στην ουσία και στον τύπο και από την νομική πτυχή. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Ε, μπορείτε όμως να θεωρήσετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, στεναρά αποφασισμένη να κάνει γρήγορα προτάσεις. Σε αυτό που επετεύχθη το τελευταίο τετραήμερο σωστά χαρακτηρίστηκε από πολλούς από εσάς ιστορική απόφαση. Με όλα τα αρνητικά που υπάρχουν σε τέτοιου είδους αποφάσεις, αλλά επειδή εγώ συμμετείχα προσωπικά για μία δεκαετία και πλέον σε τέτοιες διαπραγματεύσεις και πριν από δέκα χρόνια ε, δεν έδειξε τέτοια ταχύτητα και τέτοια αποφασιστικότητα η Ένωση στην προηγούμενη κρίση. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθύνω μια τελευταία έκκληση. Το κατανοώ και είναι απολύτως κατανοητό και το αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια ανάγκη και, δικαίωμα και το δίκαιο το έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέλει να συμμετέχει πιο εντατικά στην όλη διαδικασία λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης και στο πώς θα ε, δαπανώνται τα κονδύλια το επόμενο διάστημα. Απλώς σας παρακαλώ να γίνει αυτή η συζήτηση γρήγορα και να ληφθεί γρήγορα μια απόφαση, γιατί ε, πραγματικά ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία. Και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι όταν έχουμε αποφασίσει, έχετε αποφασίσει εσεί, χρειάζεται να αποφασίσουν και 23 εθνικά κοινοβούλια. και στη συνέχεια τα κράτη-μέλη για να προχωρήσουμε σε κύρωση. Αυτή η διαδικασία κανονικά διαρκεί πολλούς μήνες. Εδώ καλούμαστε ιδανικά να έχουμε ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια εντός του 20 για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ήδη από τις αρχές του 2021 και όχι στα μέσα ή περί τα τέλη του 2021. Και εδώ πραγματικά είναι απαραίτητη η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της ε, συζήτησης. Η επόμενη ολομέλεια τον Σεπτέμβριο αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι ζήσαμε μια ιδιαίτερη στιγμή στην ζωή του θεσμικού μας οργάνου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ε, πολιτικές ομάδες, την ε, διοίκηση του Κοινοβουλίου, τους ε, διερμηνείς. Περάσαμε μήνες πολύ δύσκολους. Κάναμε ό,τι γινόταν για να λειτουργήσει το Κοινοβούλιο. Και με την ε, λειτουργία του Κοινοβουλίου καταφέραμε να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για το οποίο οφείλω να ε, σας ευχαριστήσω για τις θυσίες ε, που έκαναν όλοι. Όλοι βεβαίως θα θέλαμε κάτι το περισσότερο, αλλά έγινε το δυνατόν με τα μέσα που είχαμε. Τώρα, η δουλειά μας συνεχίζεται και ε, βεβαίως ε, εύχομαι να ξαναβρεθούμε στο Στρασβούργο, μια από τις ε, πόλεις μας, ε, τις έδρες μας. Σας ευχαριστώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 freak oak. dag Peter.